συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Η, συνεδρία, συνεδρίαση και η ακρόαση ξεκινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον προτινόμενο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για την ακρόαση αυτή από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Κατά το τέλος εβδομάδας θα έχουμε ακρόαση και με την ε, προτινόμενη Επίτροπο Γιώροβα για θέματα δικαιοσύνης και με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Σήμερα όμως θα έχουμε ακρόαση με τον προτινόμενο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τα θέματα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων είναι ο πρώτος επίτροπος που έχει στο χαρτοφυλάκιό του τη μετανάστευση. Και νομίζω όλοι έχουμε επίγνωση της τεράστιας σημασίας αυτού του θέματος. Με βάση το παράρτημα 16 του εσωτερικού κανονισμού, που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τον προτινόμενο, τους προτινόμενους επιτρόπους με βάση τις γενικές τους ικανότητες, την ευρωπαϊκή τους αφοσίωση και την προσωπική του ανεξαρτησία θα εκτιμήσει και θα αξιολογήσει τη γνώση των χαρτοφυλακίων τους και τα επικοινωνιακά τους προσόντα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο στους προτινόμενους επιτρόπους με δύο κοινέ ερωτήσεις που έχουν συντάξει οι πρόεδροι στη διάσκεψη των πρόεδρων και τρεις ειδικέ ερωτήσεις της δικής μας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ο προτινόμενος επιτρόπος απάντησε γραπτό στο ερωτηματολόγιο αυτό και σας έχουμε μοιράσει μεταφρασμένες απαντήσεις. Η δομή τη ε, συζήτηση θα έχει ως εξή. Ο προτινόμενο επίτροπος θα κάνει μια εισαγωγική αρχική παρουσίαση το πολύ 15 λεπτών. Μετά την εισαγωγή θα έχουμε χρόνο για υποβολή 45 ερωτήσεων από τα μέλη και απαντήσεις από τον Επίτροπο. Τρία λεπτά για κάθε ερωταπάντηση. Ένα λεπτό για την ερώτηση και δύο λεπτά για την απάντηση. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων θα θέσουν ερωτήσει εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Κατά το τέλο τη ακρόαση, ο προτινόμενο επίτροπο θα έχει ένα επιπλέον πεντάλεπτο για τα τελικά του σχόλια. Λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου. Γιατί αν δεν σεβαστούμε το χρόνο μας, δεν θα περισσέψει χρόνος για να μιλήσουν όλοι και θα χρειαστεί να, δια... θα χρειαστεί να διακόπτω ε, τους ομιλητές. Έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες, οπότε ο καθένας μπορεί να μιλά και να ακούει τη μητρική του γλώσσα. Δεδομένου ότι έχουμε διερμηνία, σας θερμοπαρακαλώ να μιλάτε αργά και καθαρά. Επίσης γίνεται απευθείας αναμετάδοση της ακρόασης από το ε, διαδίκτυο και μπορείτε αργότερα να δείτε και μαγνητοσκόπηση της ακρόασης. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν θα δώσω το λόγο στον προτινόμενό μας επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο για την παρουσίασή του. Κύριε Αβραμόπουλε, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας υπενθυμίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αδιέρετες παγκόσμιες αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και φυσικά του κράτους δικαίου. Θέτει τα άτομα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, δημιουργώντας ε, την ενωσιακή υπηκότητα και δημιουργώντας μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πάνω από οτιδήποτε άλλο, η χάρτα αυτή ε, περιγράφει περί τίνος πρόκειται στην Ευρώπη που θέλουμε και καθορίζει την αποστολή που έχουμε ενώπιόν μας ε, στα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα στον τομέα αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση και σε μεγάλο βαθμό η κοινή μας υπευθυνότητα θα ελέγξει την ταχύτητα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Το γεωπολιτικό περιβάλλον εκρήγνεται. Έχουμε μια νέα απειλή τρομοκρατίας που έχει δηλώσει ότι προτίθεται να πλήξει τις κοινωνίες μας. Η ευρωπαϊκή οικονομία αγωνίζεται να βγει από την κρίση. Η ήπειρός μας ε, γίνεται όλο και γυρεότερη σε έναν κόσμο που δημογραφικά είναι όλο και νεότερος. Ε, έχουμε γκέτο στις ε, πόλεις μας που αποτελούν ε, το καλύτερο έδαφος για να αναπτυχθούν εξτρεμιστικές ιδεολογίες. Και έχουμε μορφές εγκλήματος πολύ περίπλοκες που δεν γνωρίζουν σύνορα. Και συνεχίζεται η ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορά μας που είναι οδυνηρή αντίθεση με τις κοινέ ηθικές πολιτιστικές και πολιτικές αξίες και κληρονομιά μας. Και αντιμετωπίζουμε επίσης την αυξανόμενη έλλειψη ικανοποίησης, δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να είμαι σαφής ευθύς εξ αρχής. Η απάντηση στις προκλήσεις αυτές σίγουρα δεν είναι να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη φρούριο. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα φρούρια που οικοδομήθηκαν για προστασία από εξωτερικές απειλές κατέληξαν να είναι φρούρια που έκαναν σκλάβους αυτούς που είχαν στόχο να προστατεύσουν και τελικά οδήγησαν σε απομονωτισμό. Μια τέτοια κατεύθυνση δεν είναι τμήμα της εντολής μας. Η Ευρώπη μπορεί να ευημερεί μόνο εφόσον διευκολύνει ενεργά την κινητικότητα των ιδεών, των αγαθών και των προσώπων. Η διαφάνεια και η ασφάλεια είναι πυλώνες ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτή είναι η αποστολή της ε, Επιτροπής σε σχέση με τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις. Είναι σαφής αποστολή. Πρέπει η ασφάλεια και η υποβοηθούμενη κινητικότητα να είναι βασικά συστατικά μιας Ευρώπης που θα αναπτύσσεται χωρίς φόβο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προστατεύσουμε την ταυτότητα της Ευρώπης ως ένα χώρο στον κόσμο μας που εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να εφαρμόσουμε μια ενοποιημένη και στόχο προσιλωμένη πολιτική, ούτω ώστε να προσελκύσουμε το ταλέντο και το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται κάθε κράτος μέλος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει την και θα διευκολύνει την ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας. Περαιτέρω πρέπει να εγγυηθούμε ότι το έγκλημα και η τρομοκρατία θα αποκλειστούν εκτός των εξωτερικών συνόρων και θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Κυρίες και κύριοι, για τα θέματα μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, εάν δεν κινηθούμε από κοινού ως Ένωση, δεν θα προοδεύσουμε καθόλου. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου, θα βασιστώ σε εσά, την Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών. Είμαι περήφανο που προτάθηκα ως ο πρώτος επίτροπος για θέματα μετανάστευσης. Αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση του, Προεδρε, του Προέδρου Γιούνκερ και της νέας Επιτροπής να αντιμετωπίσουν τι κρίσιμε προκλήσεις της μετανάστευση αντιμετωπίζουμε αυξανόμενο αριθμό ατόμων που επιδιώκουν προστασία εντός των συνόρων μας. Ως Ένωση που δεσμευόμεθα στην τήρηση των ε, παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ευθύνη της Ευρώπης να προσφέρει προστασία από τους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την, ε, τις διώξεις, να σεβαστούμε το δικαίωμα ασύλου και ιδιαίτερα να σεβαστούμε τη ζωή των ε, ανθρωπίνων όντων και το δικαίωμα να μην επαναπροωθούνται σε όλες τις περιστάσεις. Εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε συμβάλει ουσιοδός στην ε, δημιουργία ενός ρωμαλαίου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Τώρα έχουμε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο και η προτεραιότητά μας θα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτές τις ε, αρχές με ομοιόμορφο τρόπο. Υπάρχουν μερικοί ακόμη συμπροματικοί τομείς που πρέπει να συζητηθούν. Ιδιαίτερα η δυνατότητα να οδεύσουμε προς ένα ενιαίο καθεστώς που να ισχύει παντού στην Ένωση. Βασιζόμενοι και στα αποτελέσματα του ε, ελέγχου του συστήματος του Δουβλίνου, θα ε, αναλύσω τα ενδεχόμενα περαιτέρω βήματα. Καθημερινά ακούμε στις ειδήσει ότι φτάνουν και άλλοι μετανάστες στα σύνορά μας και ακούμε απεγνωσμένα άτομα που συχνά ε, ε, ξεκινούν ε, μοιραία ταξίδια στη Μεσόγειο. Ακόμη ένα παράδειγμα τέτοιου προβλήματος είχαμε χθες το βράδυ στην Κύπρο. Πρέπει να αυξήσουμε την δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις ασύλου, ενώ παράλληλα στηρίζουμε αυτούς, αυτούς που αντιμετωπίζουν ισχυρέ πιέσει ε, συγκυριακέ στα συστήματα ασύλου. Χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη. Και αυτό είναι δυνατό μόνο εάν τα κράτη-μέλη σέβονται και εμπιστεύονται το ένα το άλλο και αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Όμω, ε, αντιλαμβάνουμε επίση ότι η πλειονότητα των ε, μεταναστών και αυτών που χρειάζονται διεθνή προσπάθεια βρίσκονται και βρίσκουν καταφύγιο εκτός της Ένωσης από αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν ε, τις δικές τους προκλήσεις. Η διεθνής αλληλεγγύη δεν πρέπει να σταματά στα ενωσιακά σύνορα. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να στηρίξει τις χώρες ε, στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται πολλοί πρόσφυγες ή από τις χώρες ε, μετάβασης. Θα εργαστώ στενά μαζί με την συνάδελφό μου αντιπρόεδρο Μογκερίνη και τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για εξωτερικές υποθέσεις για να δημιουργήσουμε μια περισσότερο συνεκτική πολιτική για τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση. Και παράλληλα δεσμεύομαι πλήρως να ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να δεχθούν περισσότερους ε, πρόσφυγες από τρίτες χώρες. Η δυνατότητα μετεγκατάσταση των προσφύγων είναι μία από τι πιο απτέ πράξει ε, γενοδορία και αλληλεγγύη έναντι τρίτων χωρών που ε, δίνουν καταφύγιο σε πολύ μεγάλου πληθυσμού, σε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Η Ένωση πρέπει να προστατεύσει αυτού που έχουν ανάγκη, αλλά παράλληλα μπορεί να είναι αξιόπιστη αν αντιμετωπίσει την ε, παράνομη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, σεβόμενη πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όσε αιτήσει ε, απορριφθούν πρέπει ε, κατόπιν ε, οι αιτούντε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ταχαίω. Η προτεραιότητα πρέπει να είναι να του βοηθήσουμε να επιστρέψουν εθελουσίω και να του δώσουμε δυνατότητε να ενταχθούν στι χώρε όπου, από όπου προέρχονται και μάλιστα να ενισχυθούν αυτές τι δυνατότητες επανένταξης. Εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες προέλευσης, τις χώρες μετάβασης διαέλευσης και ε, επίσης όλους τους διεθνούς, διεθνείς και μη κυβερνητικού οργανισμούς. Μια σφαιρική προσέγγιση φυσικά πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση. Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη από τη διεθνή κινητικότητα, την μετανάστευση και την ένταξη. Η Ευρώπη είναι τμήμα ενός παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου πλανήτη όπου η διεθνής κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί. Πρέπει λοιπόν να αποτιμήσουμε τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, να εντοπίσουμε τις ελλείψεις που έχουμε σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Από πλευράς δεξιότητων η διεθνής, ο διεθνής ανταγωνισμός για υψηλού επίπεδου δεξιότητες είναι ήδη έντονος, αλλά η Ευρώπη χρειάζεται επίσης εργαζόμενους που θα εργάζονται σε άλλους τομείς. Θέλω να έχω τακτικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, τα κράτη-μέλη, τους επιχειρηματίες και τα συνδικάτα. Πιστεύω, μια ευρωπαϊκή ε, πλατφόρμα που να συντονίζει αυτόν τον διάλογο θα ήταν πολύ χρήσιμη. Τα πρώτα έτη εφαρμογής ε, της οδηγίας για την μπλε κάρτα κατέδειξαν, είναι αλήθεια, ότι κατέδειξαν διάφορες αρκετές ελλείψεις. Γι' αυτό ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ε, στην πρώτη φάση των δραστηριοτήτων μας στις πολιτικές του <clears throat> κατευθύνσεις γραμμές. Μία από τις προτεραιότητες μου λοιπόν θα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τους φοιτητές και ερευνητές θα καταλήξουν το 2015. Και τώρα για το Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και πρέπει να διατηρηθεί η έλλειψη ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Προπόθεση για έλλειψη τέτοιων ελέγχων είναι να υπάρχει αποτελεσματικό έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα χωρί, όπω είπα στην αρχή, η Ευρώπη να γίνει φρούριο. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο του τμήματο των εξωτερικών συνόρων που του αναλογεί. Η δυνατότητα τη Frontex πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρω για να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όμω τα μέσα που έχουν διάθεσή μα είναι επαρκή. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσουν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του Frontex και την ανάγκη και κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα πραγματικό σύστημα ευρωπαϊκών, ευρωπαίων σύνοριοφυλάκων. Η πίεση στα σύνορα και η λαθρομετανάστευση αυξάνονται συνέχεια. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε για να αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα. Ο αποτελεσματικός ε, έλεγχος και διαχείριση των σύνορων πρέπει να βασιστεί στη σύγχρονη τεχνολογία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τι δυνατότητε που μα προσφέρουν οι ψηφιακέ τεχνολογίε για τη διαχείριση τη μετανάστευση και τη κινητικότητα. Η καταπολέμηση τη εμπορία ανθρωπίνων όντων είναι προτεραιότητα. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τι ανάγκε των ανθρώπων που είναι σε απόγνωση πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και η απαράδεκτη μορφή της ε, σύγχρονης δουλείας που είναι η εμπορία ανθρώπων πρέπει επίσης να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά. Είναι λοιπόν κυρίως αυτό μία πάλι εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και στην Ένωση και διεθνώς και χρειαζόμαστε σφαιρικές απαντήσεις. Οι πολίτες μας ζητούν να τους προστατεύσουμε καθώς φοβούνται ότι απειλείται η ασφάλειά τους από την τρομοκρατία και τη βία σε καιρού σειράξεων στη γειτονιά μα και απειλών που προέρχονται από ξένου μαχητέ, χρειάζεται καλύτερα να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Το έγκλημα ταξιδεύει ανά την Ευρώπη και υπονομεύει τι κοινωνίε, αλλά και τι οικονομίε μα. Χρειαζόμαστε ένα ενημερωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή δράση που θα εστιάζει στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στι καλύτερε συνέργειε με την εξωτερική δράση. Η δράση κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος θα διευκολύνει ε, την πλήρη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η καταπολέμηση άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, η διαφθορά, θα επιτρέψει ε, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία να αξιοποιήσουν καλύτερα την εσωτερική αγορά και να αποφευθούν επίσης ε, απώλειες για τους κατοικούς προϋπολογισμούς. Αξιότιμοι κύριε βουλευτές. Ε, ε, η διατήρηση των δεδομένων είναι ένα μέσο ασφαλείας που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Τώρα έχουμε ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι θέματα προστασίας της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής και πρόσφατα έχουμε αντιμετωπίσει νέες Απειλέ από τη δρομοκρατία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών και ιδιαίτερα της σοβαρή απειλή των ξένων μαχητών. Θα πρέπει να εργαστούμε ιδιαίτερα στην πρόληψη για την καταπολέμηση ε, της ε, ακραίας ε, ε, αυτής ε, έκφανσης και του εξτρεμισμού. Η συνεργασία της αστυνομίας στην ανταλλαγή προφοριών είναι η ίδια σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής δράσης στην καταπολέμηση του εγκλήματος και εδώ ε, χωράει πολύ βελτίωση. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω την πρόθεση να συνεργαστώ στενά μαζί σας έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα. Έτσι ώστε οι πολιτικές στην Ένωση σε θέματα μετανάστευση και εσωτερικών υποθέσεων να στεφτούν με επιτυχία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε του τομεί όπου η δράση τη Ένωση μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βεβαιωθούμε ότι η δράση μα σέβεται απολύτω τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Αν με επιβεβαιώσετε, θα βοηθήσω τον εκλεγέντα πρόεδρο να χαράξει τις κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα που άμεσα συνδέονται με τη δική μου εντολή σε αυτό το σκοπό θα είμαι σε στενή συνεργασία και μόνιμη επαφή με τον συνάδελφο και αντιπρόεδρο Τίμερ μας και σε αγαστή συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν με επιβεβαιώσετε ε, θα υπηρετήσω και δεσμεύομαι γι' αυτό αυτό που μας ενώνει. Θα σέβομαι ε, με ε, απόλυτη ευλάβεια τις αρχές της Ένωσης, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις αρχές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής διαφανούς και δημοκρατικής. Θα είμαι χρήσιμος στους πολίτες χωρίς να είμαι έγκλειστος μέσα σε γραφειοκρατικά τύχη. Ταυτόχρονα θα είμαι αφοσιωμένος στις κοινέ αρχές και αξίες και θα αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα και επιμονή ε, τις νέες προκλήσεις. Επίσης, ε, σέβομαι ε, την εντολή που μας έχουν δώσει οι πολίτες. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένας χώρος ελπίδας, προόδου και ελευθερίας υπέρ όλων των πολιτών. Ε, για μένα και για μας είναι ηθική όσο και πολιτική υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you, Commissioner Designate. Ευχαριστώ κύριε υποψήφια επίτροπε για την ε, εισαγωγική σας ομιλία. Ξεπεράσατε, υπερβήκατε κατά λίγο το χρόνο σας, αλλά ε, θα το αφαιρέσω από, το τελικό σας, ε, από την τελική σας ομιλία για να είμαι δίκαιος προς όλους. Να ξεκινήσουμε τώρα τον πρώτο γύρο συζητήσεων με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, ο εκπρόσωπος και τον εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ερωτήσεις ενός λεπτού. Ο κύριος Ζομπέρτο Μετσόλα που είναι αναπληρωτής, η κυρία Μετσόλα, η αναπληρώτρια έχουμε ευρωπαϊκά θέματα που από την ίδια τους τη φύση χρειάζονται ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Πολύ συχνά μας έχουν επικρίσει, επικρίνει γιατί δεν υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Παρά τις πιέσεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αυτήν την κατεύθυνση πρόσφατα, η Ιταλία ξεκίνησε την επιχείρηση Mare Nostrum και τώρα θα ξεκινήσει και την επιχείρηση τρίτων. αλλά η επιτυχία εξαρτάται από τους πόρους που θα αποφασίσουν να χορηγήσουν τα κράτη-μέλη. Σε αυτέ τι προσπάθειε θα κάνετε εσεί ώστε να υπάρχει η σωστή επιτήρηση των συνόρων στη Μεσόγειο και να βοηθήσετε να σωθούν χιλιάδε ζωέ. Θα δεσμευτείτε συγκεκριμένα να αντιμετωπίσετε αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα ε, εμπόρων, λαθρεμπόρων ανθρώπων. Και για το άσυλο είπατε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά και υπάρχει ο βάρος επί χωρών όπως η Μάλτα, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και άλλες. Δεν θεωρείτε ότι είναι καιρός να ξαναδούμε την, ε, τον κανονισμό του Δουβλίνου. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος μηχανισμός ε, για κατανομή ευθυνών και προσφύγων μεταξύ όλων. Κύριε δύο λεπτά, κύριε Προτινόμενε Επίτροπε. Τα όλα τα θέματα μαζί και έτσι και απαντήσω σε όλα με λεπτομέρειες δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση γιατί είναι το πλαίσιο με στο οποίο φαντάζομαι θα κινηθεί το ενδιαφέρον όλων. Πρώτα απ' όλα να πούμε ξεκινώντας από το τελευταίο ότι το Δουβλίνο ε, τον τελευταίο καιρό αναθεωρήθηκε ως προς κάποιες βασικές του θέσεις. Έχουμε το άρθρο 33, έχουμε την ενίσχυση ε, της, ε, ε, ε, της, του μηχανισμού ε, κρίσεων και από την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι θα χρειαστεί να ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να γίνει μια μελέτη για να δούμε πού το Δουβλίνο χρειάζεται ενδεχομένως κάποιες αλλαγές και γιατί όχι μαζί να συνεργαστούμε για να προχωρήσουμε. Η Frontex έκανε μια πάρα και κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπω και το πρόγραμμα Mare Nostrum. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη του στο μέλλον, αλλά εκείνο μπορώ να σα πω το τρίτον έρχεται να συμπληρώσει τι δράσει τη ε, Frontex και εμεί βέβαια θα ενισχύσουμε την ε, πολιτική αυτή. Είναι επίση αλήθεια και το είπατε στην ερώτησή σα ότι δεν υπάρχουν πολλές, ε, πολλά χρήματα. Ε, αν οι πληροφορίε είναι σωστέ, αυτή τη στιγμή έχει εγκριθεί ένα ποσό 90 εκατομμύριων ευρώ και απομένουν περίπου άλλα 20 που προστίθενται. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα διεκδικήσουμε και πόρου και θα ενισχύσουμε περισσότερο τη Frontex. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε την διεθνή συνεργασία στην περιοχή. Οι χώρε που αυτή τη στιγμή υφίσταται τη μεγαλύτερη πίεση πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ του και εμεί να επιδείξουμε περισσότερο solidarity, προς, προς, περισσότερη αλληλεγγύη ε, προ ε, αυτέ. Βέβαια, Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται μια πολύ καλή μελέτη, καλή προετοιμασία και το κυριότερο μια καλή συνεργασία ε, μεταξύ μα. Γιατί, δεν σα κρύβω και ξεκινώ από αυτό, θα το πω πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση, θα χρειαστώ τη βοήθειά σα. Από μόνο του Επίτροπο μπορεί να κάνει αρκετά, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίε, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή σα θα είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν τεθεί και ως προς τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, είτε αυτό αφορά το Δουβλίνο ή την ε, Frontex, να είμαστε κοντά για να βρούμε νέους τρόπους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά, ναι έτσι είναι. Και κάτι που έχει να κάνει σχέση και, έχει σχέση με τη χώρα σας. Το relocation δοκιμάστηκε. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και αυτό βελτίωση και ενίσχυση τη αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Okay, um... Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Και τώρα, στο συγγνώμη, θα αρχίσω να σας διακόπτω, δεν λειτουργεί και το ρολόι. Περάσατε το χρόνο σας, 4 δεύτερα, όχι 32 λεπτά όπως λέει. Ε, εδώ στην Επιτροπή μας είμαστε λίγο απότομοι. Ρομπέρτα, εσύ ξεπέρασε το χρόνο σου και εσύ. Εντάξει, λοιπόν, Τώρα, συμπληρωματική ερώτηση. Ένα λεπτό. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Σίπελ. Κύριε Βραμόπουλε, σας ευχαριστώ. Μιλήσατε για την προληπτική διατήρηση προσωπικών δεδομένων, ε, την ακύρωση αυτή την οδηγία το ΔΕΚ και τόνισε ε, ότι υπάρχει ανάγκη αναλογικότητας η οποία αμφισβητείται από το δικαστήριο ε, και άλλα ευρωπαϊκά μέσα ε, βασίζονται στη μαζική διατήρηση δεδομένων και αμφισβητούνται όπως είναι ε, η ε, οδηγία για τα τραπεζικά δεδομένα και τα δεδομένα των επιβατών. Ερωτώ των αεροπορικών μεταφορών. Δεσμεύεστε ότι θα εξετάσετε κατά πόσο είναι νόμιμα όλα τα μέσα αυτά που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συλλέγουν και διατηρούν προσωπικά δεδομένα. Και δεύτερη ερώτηση, πώς θα εξασφαλίσετε στις μελλοντικές προτάσεις για ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα ποινικών διώξεων θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, η ιδιωτική ζωή και ε, άλλα συναφή. Σας ευχαριστώ κυρία Ζήπελ. Πράγματι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σαφής και για μας πλέον είναι οδηγός. Να πούμε ότι πλέον με την απόφαση του Δικαστηρίου κατέπεσε το data retention. Για όλες τις πρωτοβουλίες αναλάβουμε πλέον θα οδηγούμεθα υπό το φως της απόφασης του δικαστηρίου. Εξάλλου αυτός και είναι και ο βασικός σκοπός που καλούμεθα να υπηρετήσουμε. Θα μελετήσω, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, γιατί μου ζητάτε να δεσμευτώ, αλλά ξέρετε, οι εύκολες ε, δεσμεύσεις, ε, νομίζω σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να δείξουν και βιασύνη. Δεσμεύομαι όμως να δω αν και πώς θα μπορέσω πράγματι να έρθω σε εσά με μια νέα πρόταση. Μπορώ όμως να δεσμευτώ ότι η όποια πρόταση έλθει θα έχει όπως είπα πρωτήτερα ως αναφορά την, τον βασικό αυτό όρο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ατομικών δεδομένων και βέβαια της αρχής της αναλογικότητας. Μου είναι γνωστή σας είναι γνωστή η απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ θα έλεγα και αν σας ενδιαφέρει να μάθετε και πώς σκέφτομαι, είμαι πολύ κοντά σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και νομικής ε, εξήγησης, γιατί πιστεύω πράγματι ότι μία από τις προτεραιότητες μας είναι αυτή. Θα συνεργαστώ βέβαια με συναδέλφους, γιατί δεν είναι αποκλειστικά δική μου αρμοδιότητα, το ξέρετε αυτό, είναι ε, αρμοδιότητα και άλλων συναδέλφων, τα ε, προσωπικά δεδομένα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, έτσι ώστε από κοινού ως Κομισιόν να χαράξουμε μια ενιαία, συνεκτική, σταθερή πολιτική που θα στοχεύει σε αυτό. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς ε, και το συντονιστή, τον κύριο Τίμωθη Κέρκοπ. Ένα λεπτό. Έχω δύο ερωτήσεις, ε, κύριε Προτινόμενη Επίτροπε. Ποια είναι η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τι θα κάνει προκειμένου να αντιμετωπίσει απορρίψει νεοαφιχθέντων στα κράτη-μέλη μεταναστών. Και πώς θα εξασφαλίσετε ε, σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος του Δουβλίνου ώστε να αποφύγουμε άνθρωποι χωρίς χαρτιά, χωρίς έγγραφα και ιδιαίτερα παιδιά να διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απειλή του ISIS ε, είναι πραγματική και ε, ουσιαστική. Θέλετε το θέμα της καταπολέμησης αναχέτησης των ξένων μαχητών και το σύστημα για ένα νέο πειρα, να γίνει, όπως είπε το Συμβούλιο, προτεραιότητα στην επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Γιατί το μεγάλο αυτό πρόβλημα που έχει προκύψει με την δραστηριότητα του ISIS και με τους foreign fighters να συνιστούν πράγματι μία ε, απειλή για τις ε, κοινωνίες μας. Ε, ναι, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει μια πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος με συνέργειες και συνεργασίες ανάμεσα σε όλες τις χώρες, ώστε και με την ανταλλαγή πληροφοριών να μπορέσουμε να εντοπίζουμε τέτοιες αιστείες και βεβαίως να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Αυτό είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο είναι παράγωγο της διεθνούς τρομοκρατίας και βεβαίω φέρνει τις ε, αρχές μας πρώτης ευθύνης, τόσο τις εθνικές αρχές όσο και την Επιτροπή Πρώτης Ευθύνης να αναλάβει η μέτρα. Μου δίνει την ευκαιρία με την ερώτηση να σας πω ότι το άλλο σκέλος του χαρτοφυλακίου μου είναι βεβαίω η ασφάλεια. Αλλά η ασφάλεια δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε αυτό που είπα στην αρχή, στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ε, Ευρώπης φρουρίου. Πάντοτε, και επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτηση που με έγινε, θα πρέπει κάθε μας κίνηση, κάθε μας πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα fundamental rights, τα ε, ε, θεμελιώδη δικαιώματα ε, και τις ανάλογες αρχές. Σε ό,τι αφορά τώρα το Δουβλίνο. Απίτησα πρωτήτερα και θα το επαναλάβω. Το Δουβλίνο ως προς κάποιες πτυχές του σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε μερικά πράγματα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στη δικιά μου πρόθεση να ξεκινήσω μια τέτοια πρωτοβουλία Πρώτα πρέπει να μελετήσω, να με ενημερώσουν οι υπηρεσίε μα, να δούμε πού το Δουβλίνο χρειάζεται ενδεχομένω κάποιε βελτιώσει και γιατί όχι σε συνεργασία μαζί σα να προχωρήσουμε. Ε, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, έχω δύο δευτερόλεπτα να γυρίσω στην προηγούμενη ερώτηση γιατί δεν είπα κάτι για το PNR. Αλλά τι να κάνω, πιέζομαι από τον χρόνο. Για το PNR το συνδέω με τα data retention και έχει σημασία αυτό που σας λέω τώρα, γιατί και σε αυτό το θέμα, ενώ δουλεύει στις σχέσεις μας με την Αμερική, στο εσωτερικό της Ευρώπης πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά που προβλέπονται από την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι προστατεύονται και θα αρχίζονται τα ατομικά δικαιώματα. Thank ευχαριστώ. Σημειώνω όταν σε μερικές απαντήσεις ε, δεν έχετε εξαντλήσει το δίλεπτο, θα σας επιτρέπω στην επόμενη ερώτηση να ολοκληρώνεται. Η Σίλια Γουιξτρομ, η συντονίστρια των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε. Πριν από ένα χρόνο είχαμε το ναυάγιο έξω από τη Λαμπεντούσα. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τότε η Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν τη λύπη του λέγοντα ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να σωθούν ζωέ. Δυστυχώ έχουν μείνει κενό γράμμα όλα αυτά και κενά λόγια. Και φέτο πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Μεσόγειο, ενώ πέρυσι είχαν χάσει τη ζωή του 600 άνθρωποι. Μια και δεν υπάρχει νομικό ε, τρόπο για ε, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον άσυλο, απεγνωσμένοι άνθρωποι ε, θα ακολουθούν τέτοιες απεγνωσμένους τρόπους και οι διακινητές θα συνεχίσουν να πλουτίζουν, ενώ άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. Ο μοναδικός τρόπος ε, ε, είναι να δημιουργήσουμε ε, νόμιμους και ασφαλείς δρόμους για τους ετούντες άσυλο, για να αποφεύγουμε τέτοιες τραγωδίες. Ερωτώ λοιπόν, είστε ο πρώτος επίτροπος μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Είστε έτοιμος και πρόθυμος να υποβάλλετε προτάσεις ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς δρόμοι και νόμιμοι για τους ετούντες άσυλο. Και μέχρι σήμερα μόνο 14 χώρες μέλη ε, εφαρμόζουν ετήσια προγράμματα επανεγκατάστασης. Τι βήματα πρόκειται να κάνετε για να ενισχύσετε την κοινή πολιτική επανεγκατάστασης ώστε όλα τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέρος αυτή. αυτήν. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θα βοηθήσω περισσότερο την ερώτηση λέγοντάς σας ότι αν το σκεπτικό της ερώτησης είχε ληφθεί υπόψη κάποια χρόνια πριν, ενδεχομένω η αντιμετώπιση του προβλήματο να ήταν πιο αποτελεσματική και καλύτερη. Αναφερθήκατε στα όσα έγιναν στη Λαμπεντούζα. Το θέλησε η στιγμή τα γεγονότα της Λαμπεντούζα να συμπίπτουν με την σημερινή μου ακρόαση εδώ, γιατί ακριβώς συνέβησαν και αύριο έχουμε την επέτειο των δραματικών αυτών γεγονότων, δηλαδή στην ουσία ξεκίνησαν από σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι από σήμερα μέσα από τη συνεργασία μας μπορεί να ξεκινήσει και μια καινούργια εποχή για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Ναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Προτίθεμαι να λάβω πρωτοβουλίε. Λαμβάνοντα υπόψη και τι δικέ σα επισημάνσει, αλλά και την εμπειρία που αποκομίσαμε όλον αυτόν τον καιρό. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο, όχι μονάχα για το άσυλο, αλλά και για το, για την, ε, ε, για το irregular immigration. Πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να εφαρμοστεί η αρχή του, του, του resettlement. Και άλλες ε, ιδέες. Μπορούμε να εξετάσουμε πολλές από αυτές που θα έρθουν έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο και βέβαια να είμαστε αμήλικτοι στον πόλεμο κατά των σμάγκλες. Αυτή τη βιομηχανία, αυτό το νέο τύπο βιομηχανίας που έχει στηθεί κυρίως στο τόξο του Ευρωπαϊκού Νότου και που την ώρα που εμείς είμαστε εδώ είναι σε πλήρη εξέλιξη σχέδια. Είπατε έναν αριθμό. Επιτρέψτε να σα πω ότι ο αριθμό αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ξέρουμε πόσοι πέθαναν διότι αυτού βρήκαμε. Εκείνους που δεν βρήκαμε δεν το μάθουμε ποτέ. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να ορθώσει έναν άγχομα συγχρόνω να δημιουργήσει ένα περιβάλλον τέτοιο ασφάλεια και νομική προστασία και συγχρόνω μέσα από ιστορική συνεργασία να δούμε τρόπου ώστε να υιοθετήσουμε αρχέ νόμιμη μετανάστευση. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα μιλήσω γι' αυτό κατά τη διάρκεια τη σημερινή μα συζήτηση, εκθέτοντά σα τι απόψει μου. Πάντω, συμφωνώ με τι παρατηρήσει σα και βέβαια θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ενθαρρυντικοί προ τι χώρε για την έκδοση των humanitarian entry permits. Σα ευχαριστώ. I'm conscious that such questions require τέτοιες ερωτήσεις χρήζουν μακροσκελέστερης απάντησης, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Η κυρία Κονέλια Έρνστ έχει ένα λεπτό, είναι η συντονίστρια της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην προληπτική διατήρησή τους. Να αρχίσω ως εξή. Έχουμε την έκθεση Μωράες για τη ε, μαζική κατασκόπευση και παρακολούθηση των πολιτών στην Ευρώπη που αντιτίθεται σε αυτή. Και ζητεί η έκθεση αυτή μία αξιολόγηση ε, και αναθεώρηση ε, όλων των αντιτρομοκρατικών μέσων που έχουμε και κατά πόσο αυτά είναι συμβατά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να επανεξετάσει σε βάθος ε, τα ε, μέσα που έχουμε και μέχρι τότε να αναστείλει την συμφωνία SWIFT. Πώς το βλέπετε αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα συνεχίσετε ε, να εμένετε στην οδηγία για το PNR, για τα δεδομένα των επιβατών ή μήπως θα το ελέγξετε και αυτό κατά πόσο είναι αποδεκτό και παραδεκτό με βάση πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σας ευχαριστώ, ε, κυρία Έρνστε. εκ των πραγμάτων θα γυρίσω λίγο πίσω, συνοδεύοντας την απάντηση που σας οφείλω, με τα όσα είπα πρωτήτερα για τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά τα data retention. Ε, η απόφαση του δικαστηρίου είναι εκεί και όπως σας είπα υπό το φως, υπό το πρίσμα, το πνεύμα και τις κατευθύνσεις αυτές θα κινηθούμε στο μέλλον. Θα ήταν ευχής έργων για όλους να ολοκληρωθεί το data protection πακέτο. Είναι προϋπόθεση για όλες τις πολιτικές που πρόκειται να αναλάβουμε. Ως προς την ερώτησή σας για το SWIFT, για σχέση με την Αμερική, θα είμαι πάλι ειλικρινής μαζί σας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Γνωρίζω ότι το PNR σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Αμερική θεωρητικά λειτουργεί. Από εκεί και πέρα όμως για το εσωτερικό της Ευρώπης, εδώ είμαστε, πάντοτε υπό το φως των όσων σας είπα πρωτήτερα, να κινηθούμε υιοθετώντα νέες πολιτικές. Όταν με το καλό έρθει η ώρα να συζητήσουμε και να ψηφιστεί ένα πακέτο θα έλεγα ε, προστασίας δεδομένων, οι κανόνες αυτές θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό θα ισχύουν οριζόντια. Thank Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό από την συντονίστρια των Πρασίνων, την κυρία Σαρζαντίνη. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Κύριε Αβραμόπουλε, στις γραπτές απαντήσεις λέτε ότι χρειαζόμαστε νομικούς δρόμους για όλες ε, τις κατηγορίες εργαζομένων που ε, θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Εμείς χαιρόμαστε ως πράσινοι, γι' αυτό θα σώσουμε και ζωές γιατί όσοι περνούν τη Μεσόγειο δεν είναι μόνο πρόσφυγες, είναι και οικονομικοί μετανάστες που δεν μπόρεσαν να βρουν ένα νόμιμο δρόμο. Μπορείτε λίγο ε, να μας σχολιάσετε και να επεκταθείτε σε αυτά τα σχέδια. Πώς θα διευκολύνετε τη νόμιμη ε, είσοδο ε, για χαμηλόμισθους και με χαμηλά προσόντα εργαζομένους μη εποχιακούς ας πούμε με τις Φιλιππίνες το θέμα το γνωρίζετε, θα αντιμετωπίσετε ε, το θέμα των παρατύπων ε, ε, εργαζομένων στην Ελλάδα που μαζεύουν ελιές και έρχονται πολλές φορές από χώρες τόσο μακρινές όσο το Πακιστάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Σύριοι πρόσφυγες που έχουν οικογενειακούς δεσμούς στην Ευρώπη και χτυπούν τις πόρτες ε, των πρεσβειών μας στο Λίβανο και στην Τουρκία και τους απαντούν ότι δεν επιτρέπεται να πάτε να συναντήσετε την οικογένειά σας στην Ευρώπη. Μπορούμε να προσβλέπουμε σε εσά για τις ρυθμίσεις για την επανένωση των οικογενειών να είναι πιο προσβάσιμες για τους μετανάστες. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Ε, επιτρέψτε μου να Επιμείνω σε αυτό. Ήρθε η ώρα, ορίμασαν οι συνθήκες για να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις νόμιμης μετανάστευσης. Η πρωτοβουλία που ανέλαβε και την αναφέρατε και εσείς ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας για τους seasonal workers είναι ένα θετικό βήμα. Ακολουθεί η πρόταση κυρία Winstrom για students and researchers και βεβαίως θα προωθηθεί με σύντομους, με γρήγορους ρυθμούς και αυτό. Έχουμε την blue card η οποία βεβαίω ισχύει για high skilled εντό τη Ευρώπη, αλλά ναι, πρέπει να αποτολμήσουμε μια κίνηση προ τα εμπρός και να φτάσουμε σε αυτό που υπενηχθήκατε με την ερώτησή σα. Δηλαδή να φέρουμε στην Ευρώπη, ανάλογα με τι ανάγκε κάθε χώρα, γιατί οι χώρε είναι αυτές που ορίζουν τον αριθμό και το τι ακριβώς χρειάζονται, νόμιμη μετανάστευση. Η νόμιμη μετανάστευση, μετανάστευση είναι φράχτης για να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση και βέβαια με απόλυτο σεβασμό ε, στα ανθρώπινα δικαιώματά τους με πρώτο εκείνο των οικογενειών στις οποίες αναφερθήκατε. Η Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε βασικές θεμελιώδεις αρχές και εμείς εδώ όλοι μα όλοι, γιατί το βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, ανεξάρτητα από το που είναι ταγμένος ο καθένας, έχουμε υποχρέωση σε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που στηρίχθηκε τι αρχέ τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη τη δημοκρατία, να το σεφαρμόζουμε παντού και πάντοτε χωρίς απαραίτητα να μας το θυμίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από τη συντονίστρια της Ευρώπης της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, κυρία Λάουρα Φεράρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου ε, έβαλε οδοφράγματα, σειρματοπλέγματα στα σύνορα με την Τουρκία, είχατε πει ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία μας από τη λαθρομετανάστευση. Σήμερα το πρόγραμμα της Επιτροπής Juncker ε, φαίνεται ότι θέτει διαφορετικές αρχές ε, και θεωρεί ότι αυξάνοντα του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα θα λύσουμε το πρόβλημα. Και επικεντρωνόμαστε μόνο στου μετανάστε που θα συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Καταλάβαμε όμως ότι δεν πρόκειται έτσι να λυθεί το πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να ρηχτούν στη θάλασσα και να χάσουν τη ζωή τους ε, προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη. Πώς αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση. Δεν έχουμε μόνο την ευθύνη των ε, λαθρέα διακινητών. Είναι εύκολο να ρίχνουμε σε εκείνους μόνο την ευθύνη. Τι νόμιμη εναλλακτική λύση πρόκειται να προτείνετε εσείς, ή ενδεχομένως κάποιους ανθρωπιστικούς διαδρόμους ή τι άλλες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αποφύγουμε να εκμεταλλευόμαστε την απόγνωση των μεταναστών. Ε, αφού σα ευχαριστώ την ερώτηση, θα αναλαβει η ευρωπαικη επιτροπη ωστε να αποφυγουμε να εκμεταλλευομαστε την απογνωση των μεταναστων αφου σας ευχαριστω την ερωτηση θα να σα παρακαλέσω να μην με σπρώχνετε προς την εσωτερική πολιτική της ε, χώρας που με γνωρίζει καλύτερα. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε γενικότερα. Σε ό,τι αφορά αυτό το τείχος που χτίστηκε στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής ε, Ελλάδας, το βασικό σκεπτικό από ό,τι με να γνωρίζω δεν ήταν να αναχαιτιστεί το κύμα της παράνομης αλλά να δημιουργηθούν διεύλοι για να είναι πιο νόμιμοι οι όροι προσέγγιση στην Ελλάδα, της Ελλάδας από τη στεριά. Το αν πέτυχε ή δεν πέτυχε έχει σχετική αξία. Για κάποιους επιτυχία είναι ότι δεν έρχονται πια εκεί και πάνε στα νησιά. Για άλλου επιτυχία είναι ότι δημιουργήθηκαν νόμιμοι διεύλοι. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημά σα. Ο μόνο τρόπο είναι να δημιουργηθούν, επαναλαμβάνω, νόμιμοι όροι. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή νομοθεσία όπω την περιέγραψα πρωτήτερα, να μην την επαναλαμβάνω και σα ε, κουράζω. Το άσυλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καινούριο πακέτο τίθεται σε εφαρμογή, όπω γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του επόμενου έτου. Θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλε τι χώρε απαρέγκλητα. Και εμεί αυτή είναι η δέσμευσή μου από την στιγμή που θα κρίνεται ότι μπορώ να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα, να είμαι εκεί με τις υπηρεσίες μου και να παρακολουθώ πώς αυτό εφαρμόζεται. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε ή τις πολιτικές που πρέπει να ασκήσουμε. Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε όρους νόμιμης μετανάστευσης. Και, ε, Φεράρα, θα ήθελα να σας πω ότι ναι, μοιραζόμαστε την ίδια ευαισθησία στο πνεύμα με, τον οποίο, με το οποίο θέσατε την ε, ερώτησή σας. Αλληλεγγύη λοιπόν εσωτερική, αλληλεγγύη ε, προς τα έξω και αλληλεγγύη σε εκείνους που ζητούν άσυλο. Και όλα αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν τότε, ελήφθησαν υπό το κράτος της πίεσης που ασκήθηκε. Θα μιλήσω γι' αυτό πάλι αργότερα γιατί βλέπω αυτό το ρολόι κύριε Πρόεδρε μου κάνει τη ζωή δύσκολη εδώ. <laughs> Με έχει αγχώσει. Με κόβει το καλύτερο. Oh, το για το τέλος. Μην ανησυχείτε. Ε, και τώρα, τελευταίο σε αυτό το γύρο εκπρόσωπο των μη γεγραμμένων, ο κύριος ε, Λορέντζο Φοντάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, αυτή η επιχείρηση Mare Nostrum. Πριν από 15 μέρες ο διευθυντής της Frontex δήλωσε ότι δυστυχώς με το Μάρε Nostrum αυξήθηκαν οι αφήξεις στις Ιταλικές ακτές. Με το Mare Nostrum μήπως διευκολύναμε την κατάσταση και τη ζωή των διακινητών αντί να τους σταματήσουμε. Κατά τα άλλα διαπιστώσαμε ότι αυξήθηκαν και οι πνιγμοί μετά την επιχείρηση αυτή. Και πάντα για τη μετανάστευση θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς προτίθεστε να κάνετε μία διάκριση ε, ανάμεσα σε εκείνους που πραγματικά ζητούν άσυλο και εκείνους που έχουν κακές προθέσεις και εκμεταλλεύονται αυτή τη διαδικασία και πώς θα τους επαναπροωθήσετε αυτούς. Σε ό,τι αφορά τους ξένους μαχητές. Ακούμε ότι είναι μέχρι 3.000 οι Ευρωπαίοι που πολεμούν εκεί. Τι θα τους κάνουμε αυτούς. Θα τους αφαιρέσουμε την ηθαγένεια. Θα τους ε, απελάσουμε. Θα τους δικάσουμε. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, ξεκινώ από το τελευταίο, ότι το είπαμε και πριν, οι foreign fighters αποτελούν μια απειλή. Είπατε ότι είναι 3.000. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το νούμερο ένα από τους 3.000. Διότι είναι 3.000 ή 3.000 ή 1.500 ξέρω είναι, ξέρω όμως ότι είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Από την ώρα που ξέρουμε το νούμερο, ενδεχομένως να ξέρουμε και την ταυτότητά τους. Πάντως οι υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται Ήδη νομίζω ότι η Europol έχει ανοίξει ένα τέτοιο θέμα και ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο αυτό το επικίνδυνο για την κοινωνία μας, για την εσωτερική μας συνοχή, για την ασφάλειά μας φαινόμενο να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι preemptive way, σε ένα, με ένα προληπτικό τρόπο. Είναι μια πραγματικότητα και μας απασχολεί. Άρα είναι θέμα ασφαλείας. Για το Μάρεν Όστρουμ που είπατε, Όπω και το Mare Nostrum ήταν μια Ιταλική πρωτοβουλία, ένα Ιταλικό πρόγραμμα, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σα. Δεν ήταν τόσο αναποτελεσματικό. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι pull factor, δηλαδή ότι καθιστά το πέρασμα από, τα νότια σύνορα της ιστορίας πιο ελκυστικό για τους smugglers, αυτό να το εξετάσουμε. Εμεί παρακολουθούμε την δράση του Mare Nostrum. Διαβάζω σε εφημερίδες αλλά δεν μπορώ να το πω με τα και εμεί και εσεί διαβατευμένε, ότι υπάρχει μια σκέψη να ανασταλεί αυτό το πρόγραμμα. Η Ιταλία είναι στο τόξο που εκτείνεται η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη δραστηριότητα από smugglers και traffickers. Πρέπει να δείξουμε στην Ιταλία την αλληλεγγύη μας και να σταθούμε κοντά της η Frontex με το νέο πρόγραμμα τρίτων, το οποίο είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, μπορεί να καλύψει ενδεχομένως ένα κομμάτι της δράσης του Mare Nostrum. Ωστόσο, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις της Ιταλικής κυβέρνησης. Αλλά, επειδή πρέπει να μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια, η Ιταλία κρίνει ότι το Mare Nostrum πρέπει να σταματήσει, τότε ναι και η Ιταλία θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη αυτού του τόξου ασφάλειας του Νότου, όχι με την έννοια της security για να προχωρήσουμε σε πολιτικές ρεφουλμό. Είμαστε αντίθετοι κύριε Φοντάνα σε τέτοιες πολιτικές. Αλλά μέσα στο πνεύμα που πρέπει να κυριαρχήσει στη νέα μεταναστευτική μας πολιτική, είτε αυτό αφορά στο άσυλο στο οποίο αναφερθήκατε, είτε αυτό αφορά στο irregular immigration Πάντοτε με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκείνοι που χτυπάνε την πόρτα των συνόρων μας δεν είναι ούτε δυνητικοί τρομοκράτες, ούτε απαραίτητα παράνομα στοιχεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο που ξέρουν αυτοί καλύτερα από μας ποιος είναι και ζητούν τη φιλοξενία σε μια ευρωπαϊκή χώρα που διακρίνεται για τη δημοκρατία και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και να πω και κάτι Μια μετανάστευση για και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που όπως λέμε με γνωρίζει καλύτερα της μετανάστευσης. Όλοι είμαστε λίγο πολύ λαοί που σε κάποια στιγμή στις ιστορίες μας είχαμε μεταναστευτικά. Thank Δεν θα σας παρότρινα ε, να ε, ξεπερνάτε το χρόνο σας, ε, παρακαλώ κύριε προτιμενόμενε επίτροπε. Ας έχουμε κάποια πειθαρχία. Τώρα, ε, ξέρετε ότι τα μέλη της Επιτροπής μας είναι πάρα πολύ επιμελή και πάρα πολύ εργατικά και ε, ε, ακολουθούν τώρα τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Δίας Δεμέρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ, κάνει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας δούμε τη συνθήκη. Άρθρο 77. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαράξει πολιτική που θα έχει ως στόχο να εγγυάται τους ελέγχους των προσώπων και την αποτελεσματική επαγρύπνηση στα εξωτερικά σύνορα. Κύριε Προτινόμενη Επίτροπε, είναι γνωστές οι απειλές, οι ε, μαχητές του Ντάες και ε, οι διακινητές. Αλλά το άρθρο 77 θα πρέπει να αποκτήσει σάρκα και τα Πέντε είναι τα μέσα. Το πακέτο για τα έξυπνα σύνορα, το PNR, το SIS2, το VIS, όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα ε, και επίσης ε, πάνω απ' όλα να τροποποιηθεί ο κανονισμός Frontex. Για ποιο λόγο, διότι ευτυχώς η Frontex σώζει ζωές, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα σωστική, διότι έχει ένα κατάλογο μέσων που διαθέτει με προφορική δέσμευση, η οποία ποτέ δεν υλοποιείται. Για ποιο λόγο, διότι ο Frontex θα πρέπει να καταλάβει και εσείς επίσης κύριε Επίτροπε ότι όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις με τεράστια πίεση σε κάποιο τμήμα ή σημείο των εξωτερικών συνόρων, τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεταναστευτική πίεση. Ούτε στα χερσαία, ούτε στα θαλάσσια, ούτε στα εναέρια σύνορα. Πώς απαντάτε παρακαλώ κύριε Επιτροπέ σε αυτά τα σχόλια. Το τελευταίο ε, σημείο της ε, επισήμανσής σας και από μόνα τους, τα κράτη δεν μπορούν να κάνουν όσο θα ήθελα να κάνουν. Αναφορικά με τη Frontex. Ευθέω σα απευθύνομαι σε μια επιτροπή η οποία θα είναι ο τακτικότερο συνομιλητή μου, εάν και εφόσον κρίνετε ότι μπορώ να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα, στο μέλλον. Στηρίξτε με να ενισχύσω την Frontex. Σα το είπα πρωτήτερα, η Frontex ναι μεν υπάρχει, σε πρώτη φάση λειτουργήσε πιλωτικά, έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε και συμφωνώ μαζί σας, χρειάζεται ενίσχυση. Ενίσχυση πρώτα απ' όλα οικονομική για να καλύψει όλες εκείνες τις ειδικέ αποστολές. Τώρα ως προς το κομμάτι που λέτε και πολύ σωστά ότι δεν έχει αρμοδιότητες παρά μονάχα για την φύλαξη των συνόρων και όχι search and rescue, αυτό να το δούμε στην εξέλιξη. Και εκεί θα χρειαστεί η συνεργασία και με τα κράτη-μέλη που έχουν τις δικές τους πολιτικές. Αλλά το ότι χρειάζεται μια πιο ομοιογενοποιημένη πολιτική από όλα τα κράτη-μέλη που χρειάζονται τη βοήθεια ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει. Smart Borders. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρέπει να προχωρήσει η μελέτη, όπως ξέρετε, είναι σε εξέλιξη. Γνωρίζω ποιες είναι οι επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου και τις λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη. Και βέβαια να μην επαναληφθεί αυτό που σήμερα είναι σε εξέλιξη υπομορφή έρευνας με το SIS, δηλαδή το, ε, της και τις υπερβάσεις έξοδα. Το κόστος λοιπόν και βεβαίως το proportionality σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Σεσίλ Κέγγε. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου αφορά την πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση. Διαπίστωσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι αυτό το στοιχείο προέκυψε επανειλημμένο στη συζήτηση. Βέβαια, έχουμε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που είναι ανειδίκευτοι. Δεν είναι ούτε δικευμένοι, δεν είναι ούτε εποχιακά εργαζόμενοι, ούτε ερευνητέ, ούτε φοιτητέ. Και παρόλα αυτά θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αν θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την αρχή της ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων, και αν θέλουμε να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είπατε κι εσείς στην εισαγωγή σας, πώς προτίθεστε να θεσπίσετε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει ε, και μακροπρόθεσμα σε αυτά τα άτομα να έρθουν, να μεταναστεύσουν και που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες και παρόλα αυτά θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει καμία ευκολία, έναν σχεδιασμό και βέβαια σαφέστατους ε, κοινού κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση, το είπα και πρωτήτερα, το επαναλάβατε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη σωστή εφαρμογή των ε, υπαρχόντων ε, νομοθετημάτων και αυτό είναι μια καλή αρχή. Και βέβαια, επανέρχομαι στο πρωτήτερα, να προωθήσουμε με γρήγορους ρυθμούς την, το υποδιαπραγμάτευση students and researchers σχέδιων. Και βέβαια την αναθεώρηση της, ε, ε, της ε, Blue Card. Αυτό εξάλλου είναι και μια εντολή που μου έχει δώσει ο President-elect, ο κύριος Γιούνκερ. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης. Συνιόρα Κιουένγκε, αυτό είναι η, η απάντηση. Και νομίζω ότι η συνεργασία μας, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να έρθει η στιγμή που μαζί θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας στο να καταστήσουμε επιτέλους την μετανάστευση νόμιμη στην Ευρώπη και να φτάσουμε σε ένα πρότυπο άλλων χωρών που με ε, επιτυχία έχουν εφαρμόσει μεταναστευτικές πολιτικές και φέρουμε στην Αυστραλία ή στον Καναδά. Για να πάμε μέσα από αυτό που σας είπα πρωτήτερα στο πώς αυτές οι χώρες και είμαι σε θέση να το γνωρίζω αρκετά καλά γιατί έχω ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες ο Σάκης έχουν ανάγκη, ζητούν από άλλες χώρες να το στείλουν εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς. Όχι μονάχα σε επίπεδο διανοούμενων και πολύ μορφωμένων επιστημόνων, αλλά και για καθημερινά επαγγέλματα που βοηθούν την κοινωνία. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και προς τα εκεί θα κινηθεί κυρία Κιουέγγε η πολιτική μας και με τη βοήθεια τη δική σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιουσί Χάλα Άχο. Ευχαριστώ. Κύριε Αβραμόπολε, οι ευρωπαϊκές χώρες ήδη με μεγάλη δυσκολία ε, εντάσσουν ε, και εξειδικευμένους ε, μετανάστες, ενασμητικά προσόντα από, από τον τρίτο κόσμο. Και θα είναι μια από τις μεγαλύτερες υποκλήσεις που έχουμε να αναλάβουμε με τους ερικνωμένους προϋπολογισμούς μας. Και οι προτάσεις ε, δεν διορθώνουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί πολλής λόγος έγινε για το δικαίωμα των ανθρώπων να έρθουν στην Ευρώπη και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους μετανάστες. Δεν θα πρέπει όμως να εξετάσουμε πιο προσεκτικά και το μακροπρόθεσμο κόστος ε, και τις συνέπειες μιας αποτυχισμένης ε, κοινωνικής ένταξης και για τα κοινοτικά ταμεία και για τις κοινωνίες και τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους. Πώς βλέπετε και πού βρίσκεται την ισορροπία μεταξύ αυτών των αντιφατικών συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάτι που είναι λίγο θεωρητικό. Η, η Ευρώπη ε, χτίστηκε και συνεχίζει να χτίζεται πάνω σε διαφορετικές εθνότητες. Το απότερο όραμα εκείνων που ξεκίνησαν την προσπάθεια να ενοποιηθεί η Ευρώπη ήταν όλοι αυτοί οι λαοί, όλα αυτά τα έθνη σε κάποια στιγμή να συγκλίνουν σε συγκεκριμένε. πολιτικές. Αυτή ήταν η βαθύτερη έννοια τη ενοποίηση συμπεριλαμβανομένου και του κομματιού αυτού στο οποίο αναφέρεστε. Η Ευρώπη έχει στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια μεταναστών. Η Αμερική και η Αυστραλία είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό μεταναστευτικό οικοδόμημα. Εγώ δεν είδα σε αυτέ τι χώρε να υπάρχει πρόβλημα για την κοινωνική του ασφάλιση. Διότι αυτό είναι και ανταποδοτικό. Όταν κάποιο νόμιμα είναι σε μια χώρα κύριε αυτομάτως συμμετέχει επειδή ακριβώς είναι νόμιμα εκεί και στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με τον ασφαλιστικό του εισφορών και βεβαίως δημιουργεί. Δεν έρχεται εκεί απλώς για να δουλέψει. Δεν έρχεται απλώς για να είναι υπηρέτρια ή υπηρέτης κάποιων οικογενειών. Έρχεται για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ζητάμε να έρθουν απ' έξω εξειδικευμένοι επιστήμονες. Ναι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε, επειδή ακριβώς δείχνει και τη σολιντάριδη στην πράξη προς εκείνες τις χώρες από τις οποίες ζητάμε να μας στείλουν εξειδικευμένο προσωπικό, να μην τη στεγνώσουμε από το σημαντικό αυτό προσωπικό που θα συμβάλλει στη δική τους ανάπτυξη. Γιατί η δική τους ανάπτυξη θα αντανακλαστεί και στη δική μας εσωτερική συνοχή και πρόοδο. Θα έλεγα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Μην το φοβάστε αυτό. Άλλα πράγματα πρέπει να φοβόμαστε στην Ευρώπη. Και επειδή ακριβώς είπα στην αρχή, στο ξεκίνημά μου, ότι θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς φόβο, αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε εδώ. Um, give... ευχαριστώ. Για να δώσουμε μια αίσθηση στους συναδέλφους που βρισκόμαστε. Ε, από τις 49 ερωτήσεις, 45 είναι η 12η αυτή. Η αυτη Αναταλή Γκρισπέκ, ευχαριστώ. Κύριε ε, Προτινόμενε Επίτροπε, διάβασα τις γραπτές σας απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και σας ακούω εδώ και μία ώρα περίπου ε, την ε, πολύ εξειδικευμένη γνώση σας και τις απόψεις σας, αλλά ε, μου κάνει εντύπωση ότι δεν ακούσαμε ούτε διαβάσαμε προς το παρόν τη ε, λέξη ε, ανήλικοι, οι ανήλικοι μετανάστες. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν εσείς δεσμεύεστε για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων αυτών των παιδιών που είναι σε φάση μετανάστευσης, τι θα κάνετε για να βελτιωθεί η ιδιαίτερη κατάστασή τους και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα. Γιατί ως ανήλικοι νέοι μετανάστες είναι πιο ευάλωτοι μοιραία εξορισμού από τους ενήλικες. Ε, δεσμεύεστε ε, να υλοποιήσετε την έκθεση του Νοεμβρίου 2013 για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποια βάση και τι συνέχεια προτίθεστε να δώσετε στις παραγράφους που ζητούν και επαναλαμβάνουν το θέμα της αδυναμίας κανονικά στις δημοκρατίες μας να κρατείτε προσωρινά ή να φυλακίζετε ακόμα ένας ανήλικος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προτινέμενε. Ε, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κυρία Γκρισπέκ. Θα πρέπει να σας πω ότι η προστασία των ανηλίκων είναι υποχρέωση μας, δια νόμου, αλλά και πολιτική υποχρέωση για όλους μας. Πέρασε είμαι και είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Μπορεί να μην μπόρεσα να μιλήσω για αυτό το θέμα ακόμα, αλλά αυτό ήταν ακριβώς γιατί περίμενα να μου κάνει την ερώτηση κάποιος με τόση ευαισθησία ε, όπως εγώ. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για το 2014 θα γίνει βεβαίως σεβαστό. Και με τη δική σας υποστήριξη και τις ιδέες σας θα προωθήσουμε την προστασία των ανηλίκων. Και όχι μόνο αυτό, είναι και προσωπική μου δέσμευση. Και αν δεν το ανέφερα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εκτός του φάσματος των όσων συζητούμε. Αλλά είναι ακριβώς το πιο ευαίσθητο σημείο. Τώρα τα έχω πλέξει με τις γλώσσες. Συνεχίζω στα αγγλικά. Δεν θα πρέπει οι ανήλικοι αυτοί να κρατούνται στους ίδιους χώρους με ενηλίκους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει να φροντίσουμε τους ανηλίκους. Είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε στο μέλλον. Τα παιδιά είναι το πιο ευάλωτο και ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας μας και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στην αντιμετώπιση τους. Αυτή είναι η απάντησή μου και προσωπική μου δέσμευση πέρα από το καθήκον μου εάν με επιβεβαιώσετε ως Επίτροπο. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντική δουλειά στην καταπολέμηση της διακίνησης ανθρωπίνων όντων. Ωστόσο, εγώ ανησυχώ. Έχει φύγει από τα ανθρώπινα δικαιώματα η εστίαση και έχει περάσει την καταπολέμηση του εγκλήματος αμυγός. Παρά το ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πρωταγωνιστικό στην προστασία των θυμάτων και των δικαιωμάτων τους και στην καταπολέμηση της ζήτησης ε, το τράφικινγκ. Η μεγάλη πλειονότητα είναι γυναίκες και κορίτσια με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε πιστεύω στην ευρωπαϊκή μας δουλειά. Ερώτηση λοιπόν είστε διατεθειμένος να αλλάξετε τις προτεραιότητες σε αυτόν το τομέα και να εστιάσετε και να αντιμετωπίσετε κυρίως την καταπολέμηση του τράφικινγκ για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα ενισχύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη των θυμάτων εδώ. Το θεωρείτε τμήμα της αποστολής σας να περιορίσετε και τη ζήτηση ε, στη βιομηχανία του σεξ και τους αγοραστές αυτών των υπηρεσιών εννοώ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι προτίθεμαι να συνεχίσω και να συνεχίσω ακόμα περισσότερο την στρατηγική, την στρατηγική και τη στήριξη του Anti-Trafficking ε, Coordinator. Δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σας και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σε αυτήν την αίθουσα που διαφωνεί ότι το trafficking, αυτή η νέα ε, ε, μορφή ε, εγκλήματος, φύγει η βάναυσα και την ανθρώπινη προσωπικότητα και τη ζωή ανθρώπων. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτό το φαινόμενο της irregular ε, migration έχουμε και τους smugglers, που επιτρέψτε μου να το επαναλάβω αυτό, είναι μια βιομηχανία που έχει στηθεί κυρίως σε αυτή τη φάση των Ευρωπαϊκών Νότων, αλλά βλέπουμε με ανησυχία να εκτείνεται και προς τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και βεβαίως ο εξαπονδρισμός θα έλεγα, η εκμετάλλευση γυναικών για σεξουαλικούς σκοπούς. Εκεί υπάρχει η νομοθεσία. Και υπάρχει η νομοθεσία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, των εθνικών κρατών. Αυτό που εσείς κυρία Βιέρ λέτε και συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ομοιογενοποίηση και εναρμόνιση των πολιτικών των κρατών με βάση μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα απορρέει από τη δική μας συνεργασία. Απάντηση λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σκά Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βραμόπουλε. Αναφερθήκατε στις απώλειες ζώων που έχουμε στη Μεσόγειο και μάλιστα σήμερα ε, βλέπουμε αυτή την έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Amnesty International και που εντοπίζει το πρόβλημα στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ε, και μεταξύ των χωρών Ιταλίας, Μάλτας και άλλων και των ε, κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Τι προτίθεστε να κάνετε και πώς θα συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και να σταματήσει η άδικη αυτή απώλεια ζώων στην Μεσόγειο. Και επανέρχομαι και στο Δουβλίνο. Είπατε ότι είναι μεγάλη ευθυνή για τα κράτη-μέλη. Θα διευκολύνει την κατάσταση το να αφήσουμε τους ε, πρόσφυγες να ζητούν άσυλο εκεί που έχουν οικογενειακούς δεσμούς ή ε, όπου μιλούν τη γλώσσα της χώρας ε, αντί να ε, διακινούνται αριστερά και δεξιά. Μήπως πιστεύετε ότι αυτή θα ήταν η οπου μιλουν τη γλωσσα της χωρας αντι λύση. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά ε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, κυρία Κέλλερ, θα, να σας πω και να το επαναλάβω και μοιραία εκ των πραγμάτων θα επαναλαμβάνω κάποια πράγματα γιατί το επαναφέρουν οι ερωτήσεις που μου κάνατε ότι το πακέτο για το άσυλο είναι εκεί. Τον Ιούνιο του 2015 θα εφαρμοστεί και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που στήριξε με πάθος η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Άρα το πλαίσιο, το νομικό για το άσυλο είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί επίτευμα της συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την έρευνα και τη διάσωση. Εγώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι η έρευνα και διάσωση έχει αφαιθεί ως αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη, σίγουρα είναι καλό. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι αποτελεσματικό. Η Frontex που όπως σας είπα στην αρχή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία στην μελλοντική της μορφή και δεν αναφέρομαι στο πρόγραμμα τρίτων που έχει να κάνει με την Νότιο Ιταλία αλλά στην εξελιγμένη της μορφή και με τη συνεργασία των κρατών μελών και εκεί πρέπει να βρούμε τρόπους εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω κάποιες ιδέες αλλά μην σας κουράζω με αυτές τώρα είναι για να δοθεί περισσότερη έμφαση στο search and rescue Το, το Όστρουμ εκεί προσπάθησε να τα συνδυάσει. Αλλά όπως πολύ σωστά ελέγχθη πρωτήτερα από κάποιον εκ των συναδέλφων σας, αυτό δεν οδήγησε και στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κύριο που έχει προτεραιότητα, κυρία Κέλλερ, είναι να σώζουμε ανθρώπους. Γιατί όπως σας είπα πριν, έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία. Εγώ προσωπικά τα αμφισβητώ. Γιατί εκείνοι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να δηλωθούν για λόγους που καταλαβαίνετε θα πάρουν το, μαζί τους το μυστικό στην άλλη ζωή. Προστασία της προσωπικότητας και της ζωής των ανθρώπων. Άρα από κοινού καλούμεθα να υιοθετήσουμε μια πολιτική που να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύει και η ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κυρία Κριστίνα Βίνμπερκ. Ευχαριστώ κύριε Βραμόπουλε είναι πάρα πολύ σημαντικό το χαρτοφυλάκιο που σας εμπιστεύτηκαν και ελπίζω να το φέρετε σε πέρας αυτό το έργο. Πολλά ε, από τα ευρωπαϊκά σύνορα ε, είναι ε, περατά και στην δική σας τη χώρα. Έχουμε λάθρο μετανάστευση ε, ε, που περνούν τα σύνορα μετανάστες. Έχουμε μαχητές που επιστρέφουν από τη Συρία και από αλλού. Έχουμε συνόδευτους ανηλίκους που χρειάζονται φροντίδα και προστασία. Αυτό που μας χρειάζεται λοιπόν είναι σωστή φύλαξη των συνόρων και κυρώσεις κατά των κρατών που επιτρέπουν να διέρχεται έτσι ο κόσμος. Για να υποστηρίξουμε την νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να αποθαρρύνουμε ε, τους διακινητές και τους άλλους που εκμεταλλεύονται όλο αυτό τον κόσμο και αποκομίζουν κέρδος. Η Σουηδία κανονικά έπρεπε γεωγραφικά ε, να έχει τους λιγότερους μετανάστες ε, γιατί αυτοί θα τους αναλογούσαν. Τώρα παίρνουμε τους περισσότερους. Ε, θα χρησιμοποιήσετε το Δουβλίνο σωστά προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βίνμπεργκ. Ε, είπατε κάτι, ξεκινώ πάντοτε ανάποδα για να τα θυμάμαι και, καλύτερα, ότι η Σουηδία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ισχυρό κύμα μετανάστευσης. Πριν από πέντε χρόνια σε αυτή την αίθουσα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά θεωρούσαν ότι η regular immigration ήταν πρόβλημα μόνο του Ευρωπαϊκού Νότου. Χρειάστηκαν δηλαδή πέντε χρόνια για να γίνει αισθητό το πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ότι είναι αισθητό το πρόβλημα δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεται και από όλους με τους ίδιους όρους. Ναι, βεβαίως και χρειάζονται πιο ασφαλή σύνορα. Είναι το άλλο σκέλος της αποστολής που θα θελήσετε να αναθέσετε στον επόμενο Επίτροπο ε, Μετανάστευσης και Home Affairs των εσωτερικών Υποθέσεων. Πώς θα γίνει αυτό. Ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη μια μελέτη για το Smart Borders. Πρέπει όμως να προσέξουμε. Και το επαναλαμβάνω. Smart Borders σημαίνει χρήση νέων τεχνολογιών και διείσδυση στις, ε, στα ατομικά δεδομένα, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη για μια, όπως έχω πει, ολιστική αντιμετώπιση. Και βέβαια, η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση. Από την ώρα όμως που κάποιος καταφέρνει να έρθει στην Ευρώπη με νόμιμους τρόπους, πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να μετακινηθεί στην Ευρώπη. Και εδώ πάμε στο Δουβλίνο, στο οποίο αναφερθήκατε πρωτήτερα. Το Δουβλίνο, σας είπα και νομίζω ότι το έχετε συζητήσει πριν από μένα αυτό, σε κάποια σημεία χρειάστηκε αναθεώρηση. Δεν λέω σήμερα ότι θα το αναθεωρήσουμε. Λέω ότι θα το μελετήσουμε έτσι ώστε να εναρμονιστεί αυτή η πολιτική με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί συνολικά πλέον στην Ευρώπη και όχι μονάχα στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και βέβαια θα επανέλθω. Και μην σας συμφωνήσετε μαζί μου. Αυτή η βασική αρχή της solidarity να είναι σεβαστή από όλους, προς όλους και πρώτα απ' όλα από εμά προς τα κράτη-μέλη. Κύριε Συναδεινός. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, στο κατά τα άλλα εντυπωσιακό βιογραφικό σας μαθαίνουμε πού και τι ακριβώς διατελέσατε. Διατελέσατε παραδείγματι Υπουργό Υγεία, Τουρισμού, Εσωτερικών, Εθνική Αμήνη, Δήμαρχο Αθήνα και πολλά άλλα και εντυπωσιακά ομολογωμένο, ω τίτλοι και αξιώματα. Δεν αναγράφετε όμω τι ακριβώ επιτελέσατε, τι έχετε να επιδείξετε ω επιτυχία, ω έργο, ω κατόρθωμα. Βέβαια, επειδή όλοι μα κρινόμαστε και κρίνουμε εκ του αποτελέσματο, μάλλον δεν θα πρέπει να έχετε και πολλά να επιδείξετε ω κατόρθωμα και επιτυχία προσωπική ή και ακόμα των κυβερνήσεων που ήσασταν εξέχον μέλο. Κυβερνήσατε, κύριε Αβραμόπουλε, αλλά ξεχάσατε να υπηρετήσετε τον ελληνικό λαό. Όπω για παράδειγμα, εσκεμένα ξεχάσατε να εφαρμόσετε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία για τα αναδρομικά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αφού λοιπόν πετύχατε σε όλα αυτά, θέλετε τώρα να γίνετε επίτροπο. Και ερωτώ. Πιστεύετε ότι η συνθήκη Δουβλίνο 2 πρέπει να καταργηθεί διότι ήταν καταστροφική για τις χώρες πύλες εισόδου όπως η Ελλάδα. Συμφωνείτε και θα πείστε τους Ευρωπαίους εταίρους ότι εάν δεν δράσουμε έγκαιρα ο τεράστιος όγκος των μεταναστών αποτελεί ορολογιακή βόμβα σύγκρουσης πολιτισμών και αξιών. Ευχαριστώ. Βέβαια τα μπλέξατε λίγο, φέρατε την εσωτερική πολιτική εδώ, οι απόψεις είναι γνωστές, είναι δικές σας. Είμαι στην ελληνική πολιτική για 21 ολόκληρα χρόνια, εκλέγομαι για 21 ολόκληρα χρόνια αδιάκοπτα και είμαι περήφανος που υπηρέτησα την ελληνική δημοκρατία και το Σύνταγμα της Ελλάδος όπως εσείς για 30 χρόνια όταν είσαι στρατιωτικός. Ελπίζω να συνεχίζετε να υπερασπίζεστε τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπει το πιο, σύντομο, το πιο σύγχρονο σύνταγμα της χώρας με τον ίδιο τρόπο που το κάνατε ως στρατιωτικός να το κάνετε και ως πολιτικός. Τώρα πώς συνδέσατε τα εσωτερικά με το Δουβλίνο μια άλλη υπόθεση. Απήντησα προλίγου στους συναδέλφους σας για το Δουβλίνο και αυτή είναι η πολιτική που η κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών και δεδομένης της ε, πρόσφατης ε, νομολογίας του ΔΕΚ για, το θέμα, για την οδηγία διατήρησης των δεδομένων. Τι βήματα πρόκειται να ακολουθήσετε ώστε να εξασφαλίσετε εφαρμογή της σχετικής δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μονιστούν οι κανόνες για τη διατήρηση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της υποχρέωσής μας να εξασφαλίσουμε επαρκή ε, προστασία και ασφάλεια των πολιτών και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων αφενός και αφετέρου να έχουμε δέουσα πρόσβαση των αρμοδίων αρχών σε συγκεκριμένα δεδομένα σε περιπτώσεις καταπολέμησης σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κούντρισκα. Πρώτα απ' όλα, πολύ ορθά αναφερθήκατε στην απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ θα το πω πιο ευθέω. Το δικαστήριο σκότωσε την οδηγία και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Από και πέρα είναι εύλογο ότι θα μελετήσω αν και πώς και θα γίνει αυτό από την ώρα που κρίνεται ότι μπορώ να λάβω αυτά τα καθήκοντα θα φέρω μια νέα πρόταση. Πάντοτε όμως με άξονα, το είπα δεσμευτικά και στα εισαγωγικά μου, το επαναλαμβάνω και τώρα, του σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αρχή της αναλογικότητας. Για αυτό το θέμα όμως που θίξατε, επιτρέψτε μου να το πω, και ίσως είμαι κουραστικός, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Χρειάζεται να συνεργαστώ και με τους συναδέλφους μου επιτρόπους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αναφέρομαι στον ε, φίλο μου, αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής των κοιτήμε μας και βέβαια με την κυρία Τζούρεβα της προστασίας ε, δεδομένων. Το σημαντικότερο απ' όλα, ανοιχτός διάλογος τακτικός, συνεχής με το Κοινοβούλιο. Οι αρχές προστασίας δεδομένων είναι πολύ σημαντικές και βέβαια αυτές θα προστατεύονται με κάθε τρόπο. Μια και έχω λίγο χρόνο θα σας πω και κάτι. Όπως είπα πρωτήτερα είμαι ερετός για 21 ολόκληρα χρόνια και έχω περάσει από όλα τα στάδια όπως και πάρα πολλοί από εσά. Αυτό δηλώνει κάτι για μένα πολύ σημαντικό. Τον σεβασμό που απαιτούσα ως μέλος του Κοινοβουλίου θα τον δείχνω στο μέλλον ως Επίτροπος εφόσον εκλεγώ. Ευχαριστώ κύριος Κύρκος παρακαλώ. Κύριε Αβραμόπουλε. Μα είπατε ότι πρέπει να εκφραστεί η αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών στο ζήτημα τη υποδοχή προσφύγων. Μπορεί να μα πείτε δύο λόγια ω αξιολόγηση των επιλογών επαναπροώθηση και επανεγκατάσταση, γιατί δεν προλάβατε πριν. Επίση, μήπω να διερευνούσατε στα πλαίσια τη αλληλεγγύη, εάν σε κάποιο μελλοντικό χρόνο η εξέταση των αιτήσεων ασύλου να γίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφο, όπω για παράδειγμα είναι οι πρεσβείε σε ξένα κράτη, έστω και αν χρειάζεται αλλαγή του δικαίου σε αυτό το σημείο. Η προστασία τη ζωή προέχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Κύρκο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Κάθε μορφή ρεφουλμό, δηλαδή επαναπροώθησης, παρά την θέληση είτε εκείνου που ζητεί άσυλο ή και του regular immigrant, είναι έξω από τις σκέψεις μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίε readmission, επανεισδοχή. Κάποιες χώρες το τηρούν, κάποιες χώρες δεν το τηρούν. Πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε πρωτοβουλίε για τη σύναψη Mobility Partnership. Είναι πιο σταθερές, πιο συγκεκριμένε και πιο δεσμευτικές για τις ε, χώρες. Συνεπώς, η απάντηση στο σημείο που μου θίξετε είναι νομίζω σαφής. Το θέμα είναι ότι ξέχασα το δεύτερο σκέλος. Μπορείτε να επαναλάβει κύριε Πρόεδρε. Επανεγκατάσταση. Α, γιατί, για την ναι, επανεγκατάσταση. Ναι, γιατί, για το πού μπορεί να χορηγείται η άδεια. Πρώτα απ' όλα, εκείνοι που έρχονται στα σύνορά μα, περνάνε τι ακτέ μα και μένουν μέσα να βρουν ένα φιλόξενο περιβάλλον με σεβασμό στην προσωπικότητά του και μια και το αναφέρατε και είμαστε και οι δύο εκ των πραγμάτων Έλληνε και το συζητήσουμε. Ευτυχώ εκεί κάναμε μεγάλε προόδου και έχουμε πλέον ένα γραφείο ασύλου το οποίο ε, λειτουργεί υποδειγματικά. Αλλά και στι τρίτε χώρε. Και θα σα πω κάτι το οποίο είναι έξω ενδεχομένω στη συζήτηση και μάλιστα οι συνεργάτε μου θα μου το απαγόρευαν να σα το πω γιατί λέει πάω παραπέρα από ό,τι πρέπει, αλλά πρέπει να σα πω τη σκέψη μου. Για να γνωριστούμε και καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι όπου έχουμε σε αυτέ τι τρίτε χώρε αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φροντίσουμε να εγκατασταθεί εκεί και ένας σύμβουλος μετανάστευσης όπως συμβαίνει με την Αυστραλία, με τον Καναδά και με άλλες χώρες έτσι ώστε επιτόπου να εξετάζονται τα αιτήματα για άσυλο. Ένα μέτρο το οποίο θα εξετάσουμε πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι θα το συζητήσουμε και θα το συμφωνήσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ. The next speaker is uh, Ms. Helga Stevens. Helga. Η Helga Stevens. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε στην καταπολέμηση και αποθάρρυνση της παράνομης μετανάστευσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Είναι μια χώρα με την οποία ε, συνάψαμε πρόσφατα μια συμφωνία ε, κινητικότητας. Τι γίνεται ε, με τη συμφωνία αυτή επανεισδοχής θα εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον και σκέφτεστε να ε, προχωρήσετε σε κυρώσεις σε χώρες που δεν συνεργάζονται ε, στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες επανεισδοχής. Για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια σκέφτεστε αυτό να το συνδέσετε με τη μετανάστευση. Και επίσης, τι σκέφτεστε να κάνετε για τις διμερείς συμφωνίες. Από ό,τι φαίνεται υπολείπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Σα ε, σας ευχαριστώ κυρία Στίβεν. Σε ό,τι αφορά το Μαρόκο, πρέπει να σας πω ότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι σε εξέλιξη μια ε, έκθεση η οποία σύντομα ε, θα, μου γνωστοποιηθεί τουλάχιστον για το πώς εξελίσσεται αυτή η συμφωνία readmission που έχει υπογραφεί με το Μαρόκο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος ερωτησίας. Εάν θα επιβληθούν κυρώσεις σε χώρες που δεν σέβονται τους όρους του readmission agreement. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν είναι θέμα κυρώσεων. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα συνεννόησης μαζί τους. Τα σημεία στα οποία πάσχει η συμφωνία πρέπει πάση θυσία και των συντομότερων ετών να διορθωθούν. Εάν διορθωθούν, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε και σε ε, ε, αλλαγή πολιτικής. Τέτοιο πρόβλημα μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί. Υπάρχουν και άλλες χώρες, ξέρετε πολύ καλά, με τις οποίες έχουμε υπογράψει readmission ε, agreements, τις παρακολουθούμε και πρέπει να σας πω και κάτι εδώ. Αυτό τον καιρό που ε, γνώρισα από κοντά τις υπηρεσίες της DigiOne, θέλω να το, να το ξέρετε αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για το επίπεδο αυτών των υπηρεσιών, παρακολουθούν, κάνουν monitoring τα πάντα και δίνουν την αντικειμενικότερη και σωστότερη πληροφόρηση. Ευχαριστώ. Κυρία Χουσμενόβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αβραμόπουλε, στην γραπτή σας απάντηση δηλώνετε ότι είναι προτεραιότητά σας να κάνετε ό,τι μπορείτε έτσι ώστε η Ευρώπη να σταματήσει τις μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορά της. Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που προτίθεστε να κάνετε, ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο που έχετε ορίσει έτσι ώστε να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ενιαίο για την νόμιμη πλέον μετανάστευση. Ε, τι προτίθεστε να κάνετε, έτσι ώστε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ε, ελπίζω να μην γίνομαι κουραστικό, επαναλαμβάνοντα κάποια αυτά που είπα. Θα προτίσω να το λέω τουλάχιστον με διαφορετικά λόγια. Πρώτα απ' όλα, είπαμε εξ αρχή και είναι δεσμε, δέσμευσή μου να προωθήσουμε γρήγορου ρυθμού τι διαδικασίε για να υιοθετηθεί επιτέλους μια χάρτα νόμιμης μετανάστευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Κάτι που θα υποχρεώνει και τις χώρες να σέβονται τους κανόνες που από κοινού πρόκειται να υιοθετήσουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ήδη ένα βήμα με τους seasonal ε, workers. Νομίζω ότι οι εποχιακοί εργάτες είναι και ένα θέμα που αφορά και στη δική σας ε, χώρα. Ε, όπως επίσης και η πρόταση για τους ε, φοιτητές και τους ερευνητές. Η Blue Card επίσης είναι εκεί μονάχα που τώρα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διευρύνουμε τον, ε, το, το, πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναζητούμε ό,τι το καλύτερο διατίθεται και προσφέρεται για να έρθει στην Ευρώπη, πάντοτε κάτω από την αρχή, που όπως σας είπα πρωτήρα, να μην στεγνώσουμε τις χώρες αυτές. Παράλληλα, η πίεση θα έλεγα για την πλήρη και οριζόντια εφαρμογή της ε, αρχής του resettlement. Και βέβαια για τις χώρες στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι, solidarity. Solidarity στην πράξη. Και θα πω και κάτι παραπάνω. Σήμερα περισσότεροι solidarity έχουν ανάγκη εκ των πραγμάτων οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Αλλά όπως πολύ σωστά ελέγχθη πρωτήτερα από τη Σουηδή συναδελφό σα, το πρόβλημα πλέον έχει ξεπεράσει τον Νότο. Είναι πρόβλημα ολόκληρη της Ευρώπης. Solidarity λοιπόν συνολικά ανάμεσά μας. Και δεν ξέρουμε τι θα μας φέρουν οι καιροί και τι μας επιφυλάσσει η ιστορία για το μέλλον, όπου θα χρειαστεί να την επιδείξουμε στην πράξη. Και βέβαια και το Δουβλίνο, το επαναλαμβάνω γιατί συνέχεται άμεση μελέτη για να προχωρήσουμε αν χρειαστεί σε πιθανές βελτιώσεις. Μην ανησυχείτε για την επανάληψη, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις. κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, ακούσαμε το σχόλιο για το σειρματόπλεγμα στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας που εφάρμοσε η ελληνική κυβέρνηση, που ουσιαστικά μετατόπισε τις μεταναστευτικές ροές προς το κέντρο της Μεσογείου και κυρίως προς την Ιταλία. Η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά σας είναι η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Και είπατε ότι δεν πρόκειται να προβλέψετε νόμιμους διαδρόμους για όσους ε, βρίσκονται σε, σε κατάσταση παράτυπη αλλά ε, φεύγουν, προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους ε, από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Επιβεβαιώνεται αυτή, αυτή την προτεραιότητα. Επίσης, το Μάρτιο είχαμε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ε, θα γίνουν κάποιες προσπάθειες για την αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος του ετούντος άσυλο, ώστε να έχουμε ενίο καθεστώς για τους ετούντες άσυλο, ένα καθεστώς που θα ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτό φαίνεται στο άρθρο 78 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, ε να ξεκινήσω από το άσυλο το είπα και προτείνω και το επαναλαμβάνω, ήδη υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πακέτο για το άσυλο είναι πλέον εκεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2015. Αυτό απαντάει σίγουρα στο ερώτημά σου. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο τείχος, μούρο το είπατε, που έχει αναπτυχθεί ε, στα βόρειο-ανατολικά σύνορα της ε, χώρας που με ξέρει καλύτερα. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Ότι τότε έτσι γινόταν. Ο ευνηδιασμός τον οποίο δέχτηκαν οι χώρες μας οδήγησε την κάθε μία εξ αυτές να υιοθετήσει μία δικιά της ξεχωριστή πολιτική. Και μετά ήρθε η Ευρώπη. Και αυτό που πολύ σωστά επισημάνατε πρωτήτερα, πώς θα ομοιογενοποιήσουμε την πολιτική τη μετανάστευση. Και η απάντηση είναι μία. Νόμιμη μετανάστευση. Κανόνες. Γι' αυτό και έγινε και αναφορά στο τέλο τη ερώτησή σα στο άσυλο. Νόμιμοι λοιπόν οι κανόνε, όπω περιέγραψα πρωτήτερα. Είμαι βέβαιο ότι δεν θα αργήσει η μέρα που θα νιώσουμε όλε και όλοι υπερήφανοι σε αυτή την αίθουσα, διότι θα είμαστε αυτοί που θα αφήσουμε πίσω μα μια πολύ σημαντική κληρονομιά για το μέλλον. Μια οργανωμένη, νόμιμη μεταναστευτική πολιτική στη βάση των αρχών, των ιδεωδών και των αξιών της Ευρώπης και βεβαίω εμέσως αλλά σαφώς με οτιδήποτε έχει προκύψει ενδιάμεσα και με κορυφαία στιγμή την απόφαση όλων μας να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες αυτών των άτυχων ανθρώπων που ζουν μια καλύτερη ζωή στην φιλόξενη Ευρώπη. Uh, Ευχαριστώ. Ο Γιάννα Άλμπρεχτ είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Βραμόπουλε, κύριε προτινόμενα Επίτροπε, αναγνώρισα και χαίρομαι γιατί, για το έτσι ήταν κατηγορηματικό για την απόφαση του ΔΕΚΣ ότι αφορά την οδηγία για την διατήρηση ε, δεδομένων. Και ελπίζω να ισχύσει κάτι τέτοιο στην επεξεργασία των φακέλων και στη διαβίβαση των φακέλων επιβατών του PNR. Στο σημείο 59 της δικαστικής απόφασης, το δικαστήριο ζητά σαφή συνδεσμό μεταξύ του επιβάτη, του υποκειμένου για τον οποίο γίνεται διατήρηση των δεδομένων και τη σχέση του ε, με κάποια ε, ύποπτη ομάδα ή συγκεκριμένη περιοχή, να υπάρχουν υπόνοιες για τη διασυνδέση του με συγκεκριμένη περιοχή και φυσικά σχέση και με το χρονοδιάγραμμα ε, και τη στιγμή που ανακύπτει ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Θα αναλύσει αυτό το σημείο και θα το λάβετε υπόψη στην πρόταση αναθεώρησης οδηγία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών, το οποίο γιατί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τη συγκεκριμένη πρόταση. Το PNR εκ των πραγμάτων συνδέεται με τα ε, data retention που όπως είπαμε πρωτήτερα τα σκότωσε η απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου. Συνολικά πρέπει να το δούμε. Εγώ, αν θέλετε, δεν θα διαφωνήσω μαζί σα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι υιοθετήσουμε στο μέλλον, γιατί σίγουρα θα πρέπει να επανέλθουμε με μια νέα πρόταση με πλήρη σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, στο privacy, στην ιδιωτικότητα τη ζωή όλων των ανθρώπων. Πολλό δε μάλλον των επιβατών. Αυτό το παράδειγμα που φέρατε είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Θα πρέπει όμω να μιλήσουμε και με όλου, Να δούμε πώ μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Αν οι πληροφορίε είναι σωστέ, μόλι χτε η Ένωση Πιλότων εξέδωσε μια ανακοίνωση. Α διορθωθώ αν κάνω λάθο, αλλά ξέρετε στι εφημερίδε όταν διαβάζει κάτι πρέπει να το διπλό τσεκάρει. μια ανακοίνωση με την οποία λέει ότι όχι, μην κάνετε πίσω. Το χρειαζόμαστε το PNR και για τη δική μα ασφάλεια, βέβαια το λένε οι πιλότοι. Μπορεί όμω αυτό να οδηγήσει σε έναν ε, άλλο διαφορετικό δρόμο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη χρυσή τομή και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να συνεργαστούμε ώστε να μην ξεφύγουμε από την βασική αρχή που διέπει το πνεύμα και η απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέψει να το πω στον νιώθω θα είναι το Ευαγγέλιό μας για τα επόμενα βήματά μας. Um, Ευχαριστώ. Κυρία Τζάνις Άγνισον, ελπίζω ε, να ακούει τη φωνή μου γιατί έχω γρήπη. Η κυβέρνηση μου επισκέφθη το Καλέ και ε, για να δει πώς έχει η κατάσταση και ήμουν η μόνη Βρετανή που ε, μου εδόθη άδεια να μπω στο γραφείο του Δημάρχου. 12 εκατομμύρια στερλίνες από χρήματα των φορολογουμένων ε, θα αφιερωθούν εκεί. Ο Φιλίπ ο ε, δήμαρχος ε, ήταν πάρα πολύ έκπληκτος από την πρόταση του κυρίου Κάμερον, ε, πρόσδεκτη, αλλά τι να τα κάνω. Τον κάλεσα να έρθει να ε, γεματίσει με το UKIP και να το συζητήσει και μπορεί να προσχωρήσει και στο κόμμα, ποιος ξέρει. Τι ε, θα κάνετε για να ε, εμποδίσετε αυτό το ιδεχθές έγκλημα του τράφικινγκ και τα χρήματα που πηγαίνουν στην τρομοκρατία που είναι 15 εκατομμύρια περίπου δολάρια το χρόνο και ελεύθερη κυκλοφορία. Thank you, Mr. Mrs. Atkinson. Σας ευχαριστώ κύριε Άτκινσον. Ε, συμμερίζομαι την ε, ανησυχία σας, είναι εύλογο εξάλλου. Η ερώτησή σας σαφής. Τι κάνουμε για το trafficking, τι κάνουμε για τους smugglers, τι κάνουμε για όλους αυτούς που έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση και απροκάλυπτα και με έναν θα έλεγα προσβλητικό τρόπο ε, εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ζωή. Τώρα δεν ξέρω για το ποσό που αναφέρατε αν ανταποκρίνεται με ακρίβεια, μπορεί να είναι περισσότερο, μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ανθρώπινη ζωή ως αξία δεν ε, επιδέχεται τιμές. Θα ήθελα όμως να πω κάτι παραπάνω. Η βασική προϋπόθεση για να χτυπηθεί το smuggling είναι μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες όλων των κρατών. Και εκεί είναι το ευαίσθητο σημείο το δικό μας πώς αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε εκτροπή από τον σκοπό. Γυρνάμε δηλαδή πάλι στο ζητούμενο που είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των fundamental rights, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρακτική και αποτελεσματική λειτουργία των διοκτικών αρχών και των κρατικών αρχών. Γιατί όλοι συμφωνούμε ότι συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές. Και το παράδειγμα που εσείς βιώσατε στο Καλέ, φαντάζομαι θα το έχουν ζήσει πολλοί συμπατριώτες σας, αλλά και πολλοί που έχουν βρεθεί σε σημεία περάσματος σε άλλες χώρες, είτε λέγεται Καλέ, είτε λέγεται από την Ιταλία στην Ελλάδα ή από την Ιταλία στη Μάλτα και αλλού. Συνεπώς, ναι, η απάντηση είναι ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία για να χτυπήσουμε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο και νομίζω ότι η Europol έχει κάνει ήδη βήματα θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Συγγνώμη που σας διέκοψα προηγουμένως. Ε, φαίνεται, ε, ολοκλήρωσε, τον διέκοψε, συγγνώμη, συγγνώμη και φαίνεται ότι κουράστηκε και εγώ και πριν από λίγο αδικαιολόγητα διέκοψε και την ομιλήτρια και τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριο Κάρλος Κοέλιο. Τρει ερωτήσει για το Σέγγεν, κύριε Αβραμόπουλε. Πρώτον, 62% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν πολύ θετική την ελεύθερη διακίνηση, θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα επιτέγματα της πεντηκονταετούς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βέβαια, ε, αισθανόμαστε, έχουμε πιέσει και πολλά εσωσπαστικά κόμματα είναι κατά της ελεύθερης διακίνησης. Με ποιο τρόπο η διαφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης στον χώρο του Σέγγιν θα αποτελέσει προτεραιότητα της δικής σας θητείας. Δεύτερον, για την αξιολόγηση έχουμε ένα πραγματικό σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης που μπορεί να εντοπίσει κινδύνους στην ασφάλεια και ταυτόχρονα να τους αποτρέψει, να τους αποσοβήσει. Πώς εφαρμόσουμε το Σέγγεν, το σύστημα του Σέγγεν και τι εχέγγυα μπορείτε να δώσετε ότι θα ε, ληφθούν συγκεκριμένες και διορθωτικές δράσεις. Και τέλος, για το ΣΥΣ2, το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν Δεύτερης Γενιάς συμφωνείτε με την ε, έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, θα, το, θα λάβετε υπόψη την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Και πρόκειται για μια διαδικασία που κράτησε 6 χρόνια και στήχησε οκταπλάσια από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Κοέλιο. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσω και πάλι από εκείνο που είναι πιο κοντά σε αυτά που θυμάμαι που με ρωτήσατε. Σε ό,τι αφορά το σύστημα Σέγγεν και τους ελέγχους που έχουν γίνει. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα και πάθημα για μας και για τα smart ε, borders, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε υπέρβαση των ε, δαπανών. Και πρέπει να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό όσο ενημερώνομαι τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι τη σημασία αυτού που είπατε για το ελεγκτικό σύνολο για τους όντιτος δηλαδή που παρακολουθούν αυτό το θέμα. Το δεύτερο σημείο είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ προσωπικά μπορώ να σας ε, να σας πω και να δεσμευθώ ότι θα, θα σας ενημερώνω σε τακτικότατα χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως και, μη, και δύο φορές το χρόνο για την ε, εξέλιξη του προγράμματος Σέγγεν. Κάτι τελευταίο όμως και πιο σημαντικό. Το Σέγγεν είναι ίσως η μεγαλύτερη και πιο χειροπιαστή απόδειξη αυτού για το οποίο όλοι μαζί αγωνιζόμαστε. Για μια πιο συνεκτική, ενιαία Ευρώπη. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτό το επίτευγμα να το θέσουμε σε αμφισβήτηση. Γιατί εγώ, όπω και εσεί, διαβάζουμε σε εφημερίδε δηλώσει δεξιά και αριστερά. Εάν αύριο το πρωί με την δική σα έγκριση αναλάβω τα καθήκοντα, θα είμαι θεματοφύλακα αυστηρό ω προ την εφαρμογή του Σέγγεν και των όρων λειτουργία του. Πάντοτε ενημερώνοντα και εσά και παίρνοντα και από τη δική σας εμπειρία έτσι ώστε το σύστημα αυτό να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Και βέβαια πλήρης απαγόρευση μονομερούς επαναφοράς ελέγχων στα σύνορα χωρίς ευρωπαϊκή βεβαίωση. Thank you very much. The next speaker is... Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σιλβίγκη Γιάν, παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Οριστέντα, Επίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω, όπως και άλλοι συνάδελφοι, για τις οδούς ε, της νόμιμης μετανάστευσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να πείτε. Οπότε θα το θέσω αλλιώς. Στην γραπτή σας απάντηση λέτε ότι θα κάνετε ένα απολογισμό της ποιότητας της εφισταμένης νομοθεσίας για την νόμιμη μετανάστευση. Τι εστί αυτό και ποια ε, μέσα θα επανεξετάσετε και πώς ε, προτίθεστε να αξιολογήσετε την νομοθεσία όπως είναι η οδηγία για τους εποχικούς εργαζομένους ή την ενιαία άδεια που δεν έχει παντού μεταφερθεί όμως στην εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι σωστές οι παρατηρήσεις σας. Είπα από την αρχή και πολύ σωστά αναφερθήκατε και στην ε, ε, πρώτη μου αρχική τοποθέτηση ότι αναλαμβάνω ότι η δέσμευση να προωθήσω πολιτικές που θα οδηγήσουν μια μέρα στο να έχουμε ένα πλέγμα όρων και κανόνων νόμιμης μετανάστευσης. Μαντάμ Γιγιόν, θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου ότι η Ευρώπη δυστυχώς για όλους μας γερνάει ότι η νόμιμη μετανάστευση μπορεί να μας βοηθήσει γιατί έχουμε έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Είτε θέλουμε να το παραδεχθούμε είτε όχι είναι μια πραγματικότητα. Και βέβαια ανάγκη να ανεβάσουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας πέραν σε άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς ή και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όντως υπάρχει καινούργια νομοθεσία που είναι στη φάση της εφαρμογής της. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, και το είπα και πρωτήτερα, εκ των πραγμάτων το επαναλαμβάνω τώρα, να το δούμε πιο ολιστικά. Μέχρι τώρα το βλέπαμε αποσπασματικά. Our policy was a fragmented migration policy. Το επόμενο βήμα που θα είναι δική μας δουλειά της Επιτροπής σας, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε μια ολοκληρωμένη νόμιμη μεταναστευτική πολιτική. Και βέβαια για όλα αυτά δεν είμαστε μόνο εμεί, γιατί έχουμε να κάνουμε με την αγορά, έχουμε να κάνουμε με τα trade unions, έχουμε να κάνουμε με του ανθρώπου τη επιχειρηματικότητα και βέβαια με τη δική μα πολιτική συνεργασία. Πιστεύω λοιπόν, κυρία Γκυγιόμ, ότι τελικά εμεί θα το ζήσουμε αυτό το αποτέλεσμα και έτσι θα ξεπεράσουμε και τι ανησυχίε που προβάλλατε με το ερώτημά σα. Σα ευχαριστώ. Thank you. The next... Σας ευχαριστώ. Και τώρα, ο κύριο Φωνστός. Αξιότιμη κύριε Αβραμόπουλε, τι πιστεύετε για το άσυλο στις πρεσβείες. Αν συμφωνήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι άσυλο μπορεί αποκλειστικά να δίνεται μόνο επιτόπου και να το ζητήσουν ε, και στις πρεσβείες, τότε θα είχαμε το εξής. Ε, δεν ε, θα έχουμε πρόσφυγες στη Λαμπετούζα, δεν θα έχουν δουλειά οι διακινητές και πολύ πιο γρήγορα οι αιτήσει θα ελέγχονται επί τόπου στις πρεσβείες. Και όποιος ε, δεν μπορεί να το κάνει σε μια χώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση μπορεί να πάει στην επόμενη γειτονική ασφαλή χώρα να ζητήσει σε μια πρεσβεία άσυλο. Και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να το φέρνουμε με δικά μας έξοδα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποφασίζουμε ποιος θα τον υποδέχεται. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα λοιπόν της αίτησης ασύλου σε πρεσβείες και θα ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να υποδέχονται ε, τους ομοθρήσκους τους που διώκονται. Αυτό το γερό είναι οι χριστιανοί γνωρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, γυρνώ λίγο τη συζήτηση πίσω όταν πριν, περίπου από μία ώρα εξέφρασα και εγώ μία δική μου άποψη. Την ε, ακούσατε και εσείς και οι συναδελφοί σας ότι δηλαδή θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε για τη μεταναστευτική μας πολιτική και τις ε, υπηρεσίες εξωτερικής ε, δράσης. Γι' αυτό θα συνεννοηθώ βεβαίω με την φίλη μου την κυρία Μογκερίνη. Εγώ δεν είμαι μακριά από αυτό που εσείς είπατε. Ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να συσταθούν μέσα στα πλαίσια της νόμιμης ε, μεταναστευτικής μας πολιτικής, γιατί αυτό είναι ο στρατηγικός μας στόχος, και γραφεία στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, ιδιαίτερα σε αυτές τις τρίτες χώρες, όπου κάποιος θα μπορεί να υποβάλει το αίτημά του. Είναι μια ιδέα. Είναι μια σκέψη. Εγώ θεωρώ ότι είναι και σωστή, αν θέλετε, τη δική μου άποψη υπό την εξή Έτσι δουλεύει σήμερα η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη το να στηθεί όμως στο ευρωπαϊκό διοικητικό σύστημα και δίπλα από τις ε, αντιπροσωπείες μας εκεί. Μία τέτοια υπηρεσία χρειάζεται πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή προετοιμασία και βεβαίως αντίστοιχες υποδομές ανάλογες με τις χώρες που μπορούν να μας δώσουν την τεχνογνωσία τους με βάση την εμπειρία που αποκόμισε τα τελευταία 50 χρόνια. Συνεπώς, η απάντησή μου είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα που πρέπει να επεξεργαστούμε μαζί. Γιατί βάζει τάξη και από την άλλη μεριά δημιουργεί νόμιμους τρόπους για να μπορούν να υποβάλλονται τα αιτήματα. Το τι θα αποφασίζει η Ευρώπη είναι άλλη υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ τη μεταναστευτική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Η, ερώτηση υπερθυμών 27 από τον κύριο Λουί Μισελ. Κύριε Προτινόμενο Επιτροπέ, για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία με αυστηρό σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είπατε ότι αυτό είναι στόχος. Θέλετε με ανθρώπινο τρόπο να ασχοληθείτε με τα θέματα των μεταναστών, ε, με σεβασμό επίσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μεγάλη ρητορική δυνότητα υπέρ της διατράνωσης των γενικών οικουμενικών αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ όμως για να ε, βεβαιωθώ θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις θα πραγματοποιήσετε μελέτη ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών και τη ενωσιακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και το κατά πόσο οι νομοθεσίε αυτέ συνάδουν με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί στην έκθεσή μου για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 2015 είχα θέσει σχετικό αίτημα. Και δεύτερη ερώτηση γιατί δεν ικανοποιήθηκα πλήρως από μια προηγούμενη απάντηση. Πώς θα εξασφαλίσετε τον αυστηρό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των άσυλων από τα κράτη-μέλη από τη στιγμή που θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είπατε κάπως αφηρημένα, ε, είπατε, μιλήσατε με, με κάποια σάβια ε, ε, για την δημιουργία φραχτών στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Ε, και μέχρι στιγμής ε, είχα κάπως καθησυχαστεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποφύγατε την ε, ερώτηση, που κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ σημαντική, γιατί τα σειρματοπλέγατα δεν είναι ανοιχτή Ευρώπη, σε καμία περίπτωση δεν είναι Ευρώπη των αξιών. Σας θέτω λοιπόν ευθέως την ερώτηση. Τι γίνεται με τις φράχτες αυτές και τα σύρματοπλέγματα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Θα ήθελα να με καθησυχάσετε λοιπόν. Ευχαριστώ με ε, Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να, θα ήθελα να σας πω κάτι, κάτι γνώμη σημαντικό. Προλίγου. Δεν ρωτήθηκα για τη δική μου άποψη για τους φράχτες. Δεν, δεν ρωτήθηκα εγώ τι πιστεύω για τους φράχτες. Έδωσα εξήγηση για ποιο λόγο έγιναν αυτά. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, αν και έχω απαντήσει με τις αρχικές παρατηρήσεις, είμαι εναντίον οποιοδήποτε μέτρου που θα κατασύσει την Ευρώπη φρούριο. Και μάλιστα το εξήγησα. Λέω θα οδηγηθούμε σε isolationism, δηλαδή σε απομονωτισμό. Εγώ πιστεύω σε μια ανοιχτή, ελεύθερη, δημοκρατική Ευρώπη. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Διότι μια Ευρώπη χωρίς σύνορα είναι σαν να λέμε ένα κράτος χωρίς σύνορα έτσι ώστε όλα να λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και με βάση αυτό που είναι και δική σας ευαισθησία και έχετε αγωνιστεί για αυτό, δηλαδή το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις ανθρώπινες ελευθερίες και στα προσωπικά δεδομένα. Θα ήταν ευχής έργων να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν το Data Protection Package. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, εάν και εφόσον προτίθεμε, γιατί πρέπει να πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, εσείς μου δίνετε την ιδέα τώρα για την ανάλυση της, των εθνικών νομοθεσιών, η απάντησή μου είναι, ναι. Και για να πω και κάτι παραπάνω, για να σας βοηθήσω, αν το είχατε πει και παλιότερα, απορώ πως και δεν έχει γίνει τώρα. Γιατί για να φτάσουμε σε μια ομοιογενοποιημένη, εναρμονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική, πρέπει να ξέρουμε πώς σκέπτεται, ποιες είναι οι απόψεις και ποιο είναι το θεσμικό σύστημα κάθε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν απαντώ στο ερώτημά σα με ακρίβεια και λέω ναι και σα ευχαριστώ για την ιδέα που μου δώσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Χρυσόγωνος, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, το άρθρο 15 της Οδηγίας 115 του 2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ως ανώτατο όριο κράτησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών τους 18 μήνες. Ωστόσο, με τη γνωμοδότηση 44 του έτους 2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία επικυρώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, συνάδελφό σας στην ελληνική κυβέρνηση, έγινε δεκτό πως σε περίπτωση κράτησης αλλοδαπού επί 18 συνολικά μήνες κατόπιν προηγούμενης απόφασης απέλασής του, τα αρμόδια όργανα δύνανται, να επιβάλλουν σε αυτόν το μέτρο, ακούστε, της υποχρεωτικής διαμονής στο χώρο κράτησης χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, επαόριστον. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμφωνία ή μη της πρακτικής αυτής των ελληνικών κρατικών αρχών προς το ενωσιακό δίκαιο και πώς σκοπεύετε να δράσετε αν και άλλα κράτη-μέλη στο μέλλον ενθουσιαστούν και ακολουθήσουν παρόμοιες πρακτικές. Ευχαριστώ κύριε Χρυσόγονε. Δεν νομίζω ότι το ρήμα ενθουσιάζομαι πηγαίνει σε αυτή την περίπτωση γιατί ακόμα και αν συμβεί αυτό δεν νομίζω ότι το κράτη, τα κράτη τα κάνουν με ενθουσιασμό. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της Ελλάδος. Λέω από την αρχή ότι η πρόθεσή μου από την ώρα που κρίνει το Κοινοβούλιο ότι μπορώ να λάβω αυτή τη θέση δεν θα είμαι εδώ ως Έλληνας υπουργό. Τυχαίνει να έχω την ιδιότητα αυτή ακόμα, αλλά δεν μιλάω με αυτήν την ιδιότητα. Γι' αυτό και θα είμαι και πολύ ειλικρινής και σαφής και ευθύ στην απάντηση. Κράτηση μεταναστών πάνω από 18 μήνες απαγορεύεται. Γνωρίζετε όμως, γιατί είστε ένας εκ των πλέον διακεκριμένων Ελλήνων νομικών και συνταγματολόγων, ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι, γνωμο, είναι γνωμοτικού χαρακτήρα. Δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα. Είπατε ότι το δέχτηκε κάποιος υπουργό. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ανεξάρτητα αν το δέχτηκε το δέχτηκε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ. Και πρέπει να το εξετάσουμε με άμεσο διάλογο μιλάω πλέον από την πλευρά τη Επιτροπή, με τι ελληνικέ αρχέ. Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Ξόγωνε, και το υπονοείτε μέσα από την ε, ε, ερώτησή σας, δεν είναι εγκληματίες. Αλλά μετά το 18 μηνό του πρέπει να μπουν μέσα στην παραγωγή. Προσέξτε όμω. Έχουμε δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη μια γκρίζα ζώνη. Και η γκρίζα ζώνη ενέχει ένα κίνδυνο για του τους Να είναι περισσότερο εκμεταλλεύσιμοι επειδή ακριβώς είναι undocumented, κυκλοφορούν μέσα στις κοινωνίες μας και κάποιοι επιτίδιοι μπορούν να τους εκμεταλλευτούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την κρίζα ζώνη πρέπει να την τελειώνουμε. Και ο μόνος τρόπος είναι αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη σήμερα, η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων νόμιμης μετανάστευσης. Και το πακέτο του ασύλου απαντάει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα από την ώρα που θα εφαρμοστεί από τον επόμενο Ιούνιο. Η κυρία Εύα Ζωλή, παρακαλώ. Κύριε οριστέντε Επίτροπε, η Πολωνία ε, αναγνωρίστηκε ότι συμμετείχε και ε, ήταν συνένοχος με τις ε, δραστηριότητες και τα προγράμματα της ε, CIA, όπως και άλλες εννέα χώρες. Έχει τεκμηριωθεί και έχει αναγνωριστεί αυτό πλέον. Εσείς πώς προτίθεστε να συνεισφέρετε ε, στην ε, καταπολέμηση της ατιμορρησίας, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επειδή συμμετείχαν στις παράνομες παραδόσεις, παράνομες κρατήσεις, όσο και βασανιστήρια ανθρώπων που υποπτευόταν η CIA για τρομοκρατία προτίθεστε να παρακολουθήσετε και να δώσετε συνέχεια στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτά τα προγράμματα. Και αν ναι, με ποιο τρόπο θα βοηθούσατε τα κράτη-μέλη να κάνουν γρήγορες έρευνες όσο και ανεξάρτητες και σε βάθος για όλους τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες για απάνθρωπη και ε, ταπεινωτική συμπεριφορά όσο και βασανιστήρια ε, στα οποία εκείνα ήταν συνένοχοι ε, είτε με τη σιωπή τους στα πλήσια δραστηριοτήτων της CIA. Ξεκινώ λέγοντάς σας ότι απάνθρωποι ταπεινωτική, προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συμπεριφορά είναι ασυγχώρητη από όπου και αν προέρχεται. Πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτήν την έκθεση ε, δεν τη γνωρίζω σε βάθος. Ανεξάρτητα όμως αν τη γνωρίζω ή δεν τη γνωρίζω, η ερώτησή σας δεν έχει να κάνει με το θέμα αυτό, αλλά με το ποιε είναι οι βασικές δικές μας αρχές. Η Ευρώπη στηρίζει την ύπαρξή της σε μια θεμελιώδη αρχή, πέραν των άλλων, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και εδώ δεν κάνει κανένα διαχωρισμό. Και επειδή έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου για την μετανάστευση και για τα Home όπου εκεί ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την ασφάλεια, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι και εκεί ως εκ του χρέους και του καθήκοντός μου θεματοφύλακας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και αυτές ήταν οι οδηγίες που θα δοθούν στις υπηρεσίες του αυριανού Επιτρόπου, εφόσον κρίνεται ότι μπορώ να είμαι εγώ, γιατί έτσι θα λειτουργούν. Και η Ευρώπη της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι η μεγάλη κατάκτηση και αυτό πρέπει να καλλιεργούμε και σε αυτό το χώρο, αλλά και κυρίως μέσα από τα μέτρα και τις πολιτικές που υιοθετούμε. Γιατί η Ευρώπη πάνω απ' όλα είναι πολιτισμός. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ιγνάτσιο Κοράο. Κύριε Αβραμόπουλε, άκουσα με προσοχή τις ερωτήσεις που σας έθεσαν οι συνάδελφοι και άκουσα και τις δικές σας απαντήσεις. Είστε παλέμαχος πολιτικός και χρησιμοποίησατε την πλούσια πείρα που έχετε ε, για να δώσετε μια πολύ καλή εικόνα. Τώρα, έχω ερωτήσεις συγκεκριμένες για τον ε, κανονισμό του Δουβλίνου και τους ετούντες άσυλο θα πρέπει να έχουμε ισότιμη κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κατά τη γνώμη μου. Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία σχετικά. Και μία πιο προσωπική ερώτηση. Στο διαδίκτυο ε, βλέπουμε, βλέπουμε μία φωτογραφία σας ε, με ε, ένα όπλο που κρατάτε στον ώμο σας κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Κοντά σε αυτό το φράχτη με το σειρματόπλεγμα. Είναι πραγματική η φωτογραφία, γιατί αν δεν είναι φωτομοντάζ είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη η εικόνα και είναι σαν να βάζουμε το λίγο, το λίγο να, φυτά, να φυλάει τα πρόβατα, αν είναι όντως αληθινή αυτή η φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα, να σας πω αυτή τη φωτογραφία την είδα και εγώ. Και μάλιστα η φωτογραφία με έχει σε ένα κέντρο εκπαιδεύσεως στην Τρίπολη, που είναι δίπλα από το χωριό της μητέρας μου στην Αρκαδία, όπου εκπαιδεύονται εκεί οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες. Και επειδή εγώ δεν πηγαίνω στις ορκομοσίες τους για το Θεό Αθήνα και τις τελετές, αλλά και θέλω να δω ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπαιδεύονται οι Έλληνες στρατιώτες. Όταν βρέθηκα κοντά τους, βεβαίως και πήρα στα χέρια μου το όπλο. Μην νομίζετε ότι είμαι φίλος των ε, όπλων. Εξάλλου το χειρότερο πράγμα είναι να έχεις όπλο και να μην ξέρεις και να το χρησιμοποιήσεις. Συνεπώς αυτή η φωτογραφία ήταν μια φωτογραφία χιουμοριστική, την οποία έβαλε ένα περιοδικό. Και βέβαια ποτέ, μα ποτέ δεν θα έκανα μία επίδειξη στα σύνορα με την Τουρκία. Και επειδή προφανώ το γνωρίζετε, πρέπει να ξέρετε ότι είμαι ο αρχιτέκτονα τη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ω Δήμαρχο Αθηναίων το 1995 είχα ανοίξει τι πόρτε για σχέσει ανάμεσα στου λαού και αυτό έγινε case study και έγινε endorsed στα Ηνωμένα Έθνη, έθνη κάτω από τον τίτλο Cities Diplomacy. Γιατί πιστεύω στη συνεργασία των λαών και όπω μου είχε πει τότε ο Κόφι ήρθε η ώρα να χτίζουμε την ειρήνη από τον από τα κάτω προς τα πάνω. Άρα μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις. Αλλά το χιούμορ χιούμορ. Και θέλω να σας πω ότι στο γραφείο μου αν έρθετε θέλετε πάρα πολλές καρικατούρες. Μάλιστα λέω ότι όσο περισσότερες καρικατούρες μου κάνουν τόσο περισσότερο θα υπάρχω στην πολιτική. Τώρα σε ό,τι αφορά την ισότιμη κατανομή. Κάθε χώρα έχει τις ανάγκες της. Αυτό είναι. Κάθε χώρα θα κρίνει πόσοι θα πάνε στη, στην χώρα αυτή. Τι χρειάζεται. Επιστήμονες, εργάτες, ταξιτζίδες, κομμότριες, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να χρειαστεί. Η κεντρική όμως η μεταναστική πολιτική από την ώρα που είναι νόμιμη θα κάνει την κατανομή. Άρα δεν είναι αναλογικό, είναι σύμφωνα με τις ανάγκες. Φτάνει να είναι νόμιμο. Κύριε Ρασιντάντα, τι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Προτινόμενε Επίτροπε έγινε λόγος για συμφωνίες με τρίτες χώρες για την κινητικότητα για να οργανωθεί βεβαίως η νόμιμη μετανάστευση με τη δική τους δέσμευση να ε, βοηθήσουν στην καταπολέμηση της λαφρομετανάστευσης και την ε, εγκληματικότητα που συνδέεται. Πώς θα φροντίσετε λοιπόν να εφαρμόζονται σωστά και να εκτελούνται αυτές οι συμφωνίες. Γιατί δεν μας απάντησε ποτέ ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως οικονομικοί πόροι που δίδονται στα πλαίσια αυτών των εταιρικών σχέσεων, πώς θα δαπανώνται και πέρα από τη μετανάστευση, νόμιμη και παράτυπη, ε, αυτή φέρνει και την κινητικότητα και τη μεταφορά του οργανωμένου εγκλήματος κάθε είδους. Διακίνηση ανθρώπων, πορνεία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ποιες είναι οι υπόλοιπες τρίτες χώρες που θα συνάψουμε συμφωνίες μαζί τους και πώς θα τις φέρετε ενώπιον των ευθυνών τους για να αντιμετωπίζουν ε, αυτά τα εγκληματικά δίκτυα αποτελεσματικά. Και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε σε αυτά ως βιομηχανία. Ερώτησε και η κυρία Στέβενς, αλλά δεν ξέρω αν απαντήθηκε πραγματικά για τις κυρώσεις κατά των τρίτων αυτών χωρών. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω απήντησα και για τις ε, ε, ε κυρώσεις. Εφόσον με αυτές τις χώρες έχουμε υπογράψει ε, συμφωνίες για readmission ή ακόμα και mobility partnership. Αλλά πέραν αυτού θέλω να σας πω ότι ναι, πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλες αυτές τις χώρες πρόθεσή μου είναι να προωθήσουμε τέτοιες ε, συμφωνίες. Και μια και με ρωτήσατε με ποιες χώρες, αλλά ξεκάθαρο αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε καταρχήν με τις ε, χώρες ε, της ζώνης της Βορείου Αφρικής. Κάποιες από αυτές είναι σε θέση να το κάνουν, κάποιες άλλες όμως περνάνε δύσκολες στιγμές. πούμε με τη Λιβύη, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βρέθηκα στη Λιβύη πριν από λιγου μήνε και δεν σα κρύβω ότι ήταν από τι λίγε φορέ τη ζωή μου που φοβήθηκα. Η κατάσταση είναι χαοτική. Δεν μπορεί να βρει συνομιλητή αυτή τη στιγμή στη Λιβύη αλλά πρέπει να τι προτάξουμε ως χώρες με τις οποίες μπορούμε να συνοηθούμε. Βεβαίως, αμήλικτο πόλεμος κατά του smuggling και του trafficking. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι που υπενηχθήκατε, διαφάνεια, transparency, σε όλα αυτά. Χρηματοδότηση, έλεγχο, διαφάνειας και accountability. Δηλαδή πρέπει η Επιτροπή σα να δέχεται συχνά και να υποβάλει και αιτήματα πέραν των πρωτοβουλίων που θα πάρουμε εμείς για να έχετε πλήρη εικόνα όλα αυτά τα ποσά που διατίθενται, πού πηγαίνουν και αν υπάρχει ανταποδοτικότητα στην, στην ε, πράξη. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, το θυμίζω αυτό, για το 2015 κατά του smuggling. Το συμπέρασμα είναι ότι ναι, πρέπει να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια, θα με επιτρέψετε να θυμίσω και μια ακόμα φορά ότι γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία και με την κυρία Μογκερίνη, η οποία έχει την ευθύνη της εξωτερικής δράσεως, γιατί όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πακέτο σχέσεων με άλλες ε, χώρες και δεν προτίθεμαι σαν παλιές διπλωμάτης να κάνω το λάθος να υπερβώ τα πλαίσια των δικών μου δικαιοδοσιών. Κυρία Μίριαμ Ντάλι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προτινόμενα Επίτροπε. Πολλές φορές και σήμερα ακόμη ακούσαμε πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της Frontex και εκφράσα την επιθυμία για την ενίσχυση της Frontex και μάλιστα στη δική μας υποστήριξη για να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τη Frontex. Η Frontex επίσης ετοιμάζεται να συντονίσει μια νέα επιχείρηση, το πρόγραμμα Τρίτων. Μας είπατε ότι το πρόγραμμα Τρίτων, η επιχείρηση Τρίτων θα βοηθήσει τη Frontex και θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα τρίτων στον έλεγχο των συνόρων, στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Μας είπατε ότι η Frontex έχει την αρμοδιότητα να ενισχύσει τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα για έρευνα και διάσωση. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τι μέτρα τελικά θα λάβετε ώστε αυτοί οι απεγνωσμένοι άνθρωποι που χρειάζονται κατεπηγόντως τη βοήθειά μας θα τύχουν διάσωσης. Ναι, πολύ σωστά ε, ε, αναφερθήκατε σε αυτό που είπα πρωτήτερα για την, ε, για την Frontex. το mandate της Frontex, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν είναι να, να έχει την ευθύνη του search and rescue. Το κάνει συμπληρωματικά. Γνωρίζετε πολύ καλά το δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει σε κάθε πλοίο, πολλό δε μάλλον στα ε, σκάφη της Frontex, ο Τσάκης προκύπτει ανάγκη να συνεισφέρουν στη διάσωση ζών. Και θα πω κάτι, από το ρέκορντ μέχρι στιγμής της Frontex έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου η Frontex έσωσε ζωή. Αλλά, ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι η βασική της αποστολή. Είπα πρωτήτερα και το επαναλαμβάνω ότι πρόθεσή μου είναι, εφόσον αναλάβω αυτά τα καθήκοντα, να αναλάβω πρωτοβουλίε για την ενίσχυση τη Frontex. Όχι μονάχα για το τόξο του Ευρωπαϊκού Νότου. Ε, δεν ξέρουμε πού αλλού μπορεί να προκύψει ανάγκη. Σήμερα ξέρετε ότι είναι σε ανάπτυξη επτά προγράμματα της Frontex. Τρία στο Αιγαίο, δύο στην Νότια Ιταλία και τρία κοντά στην Ισπανία. Η Frontex δεν έχει όμως επάρκεια. Ούτε σε μέσα, ούτε σε δυνατότητες και βέβαια δεν έχει την απαραίτητη οικονομική στήριξη συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, αλλά η βασική της αποστολή είναι η προστασία των συνόρων. Όταν λοιπόν λέμε για ενίσχυση της Frontex, δεν θα αργήσει η μέρα που θα έρθει εδώ ενδεχομένω μια πρόταση για να δούμε μήπως τις αναβαθμίσουμε και το ρόλο συμπεριλαμβάνοντας και το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε πρώτα. Εγώ προσωπικά, γιατί πρέπει να, από την ώρα που έχετε μπροστά σας κάποιον που θα επιλέξετε ή όχι να λάβετε τα καθήκοντα, να ξέρετε και πώ σκέπτεται και ο ίδιο. Μην κρύβουμε δηλαδή και τι σκέψει μα. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι η Frontex πρέπει να εξελιχθεί και με το ενισχυμένο πρόγραμμα τρίτων, το οποίο είναι συμπληρωματικό και θα το δείτε να λειτουργεί στην πράξη στην ε, περιοχή της ε, Ιταλία, να εξελιχθεί σε ένα όργανο το οποίο θα σώζει ζωέ συγχρόνω όμω θα προστατεύει και τα σύνορα. Προϋπόθεση όμως αυτά που σας είπα πρωτήτερα. Και για όλα αυτά δεν θα αργήσει η μέρα που θα τα συζητήσουμε σε αυτήν την αίθουσα και πάλι. Ο κύριος Μίχαου Ουγιασδόφσκι. Η ερώτησή μου αφορά ακριβώς αυτό το εμπόριο ανθρώπων για το οποίο μιλήσαμε Πώς κρίνετε την οδηγία του 2011. Κατά τη γνώμη σας η οδηγία αυτή εφαρμόστηκε αποτελεσματικά από τα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το, το ύψος των τιμών, την αυστηρότητα των τιμών και την κατάσχεση των εργαλείων του, ή των μέσων του εγκλήματος. Πώς κρίνετε αυτή την οδηγία από το 2011 και σκοπεύετε να αναλάβετε ε, ως αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα αυτά κάποια μέτρα για νομοθετικές αλλαγές για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα ήθελα να μας αξιολογήσετε συγκεκριμένα αυτή την οδηγία του 2011 και ποιες ενδεχομένως νομοθετικές αλλαγές θα προτείνετε. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ ενημερώθηκα για αυτήν την ε, οδηγία και πρέπει να σας πω ότι η πρώτη εκτίμηση που μπορώ να κάνω, αν και δεν έχω αυτήν την ευθύνη αυτήν την ώρα, είναι ότι σίγουρα παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις. Δεν πάβει όμως από το να κινείται στη σωστή ε, κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η ενίσχυσή της είναι μια πολύ σωστή ιδέα. Δεν μπορώ όμως από τώρα να σας πω προς ποιαν κατεύθυνση. Και τούτο διότι όταν με το καλό και εφόσον εσείς κρίνετε αν λάβετε τα καθήκοντα θα ζητήσω πληρέστερη ενημέρωση. Η πρώτη καταρχήν όμως που έχω είναι ότι είναι μια σωστή οδηγία που ως προς την εφαρμογή της παρουσίασε κάποιες ελλείψεις τις οποίες και πρέπει να βελτιώσουμε. Πίτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενε Επίτρεπε, στην επιστολή που σας απίφθινε ο κύριος Γιούνκερ λέγει ότι η Ευρώπη θα πρέπει καλύτερα να διαχειρίζεται τη μετανάστευση σε όλες τις πτυχές της. Φοβούμαι όμως ότι θα συμφωνούσαν και δικοί μου ψηφοφόροι ότι υπάρχει ανησυχία για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και θα πρέπει ε, να δικαιολογήσουμε και τη δράση μας και τις αρχές και τις αξίες μας, στις οποίες και εσείς αναφερθήκατε. Έχω δύο ερωτήσεις. Τι προτίθεστε να κάνετε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να βελτιώσετε την ε, ένταξη των μεταναστών προς όφελος όλων και πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε αλλά και να επηρεάσετε τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για αυτό το θέμα. Διότι εάν κόμματα ε, που έχουν ε, σημαία τους ε, την μετανάστευση και αρχίζουν και φτάνουν στις κυβερνήσεις, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε Γέζεκ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που εκμεταλλεύονται την φτώχεια, την οικονομική κρίση, την ανέχεια, την εξαθλίωση. Και πάνω εκεί χτίζουν τις δικές τους προτάσεις έχοντας ως εργαλείο το λαϊκισμό που είναι μία από τις χειρότερες μορφές πολιτικής. Είναι ένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι όταν σταδιακά αρχίζουν να ξεπερνούνται οι λόγοι που το έχουν προκαλέσει και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας, την οικονομική κρίση, της Ευρώπης ενώ την οικονομική κρίση, αλλά και εξωτερικά τις μεγάλες απειλές και την κλιμακούμενη κρίση σε ζώνες υψηλής ανασφάλειας, όπως είναι η Μέση Ανατολή ή ακόμα και το τόξο αυτό που εκτείνεται από την Τινησία μέχρι την Ουκρανία, όλα αυτά θα αρχίσουν να περιορίζονται. Και τούτο γιατί. Διότι η κουλτούρα των λαών της Ευρώπης είναι βαθιά δημοκρατική. Η Ευρώπη έχει υποφέρει στο παρελθόν από δικτατορίες, φασισμούς, που την οδήγησαν σε μεγάλες περιπέτειες και αυτό είναι μέσα στο DNA των λαών. Απλώς κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν μέλλον στην Ευρώπη και σας μιλώ αυστηρά με πολιτικούς όρους. Από εμά εξορτή. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό που λέτε είναι η Ευρώπη. Η λύση είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη της αλληλεγγύης και βέβαια μέσα από τις πολιτικές που μέχρι στιγμής τουλάχιστον στη συζήτησή μας έχουμε περιγράψει, δηλαδή η στήριξη των βασικών αξιών πάνω στις οποίες έχουμε θεμελιώσει το ευρωπαϊκό οικοδόμα. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί τη μεγάλη ευθύνη όλων μας ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο καθένας ή καθεμιά από εμά είτε στα όργανα της Ευρώπης είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στα Εθνικά ε, Κοινοβούλια. Αυτή είναι η απάντησή μου, η γενική, με κάποιες σαφέστατες επισημάνσεις για τους κινδύνους, που όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο ισχυρές ώστε να μας φοβίζουν. Η δημοκρατία και η δημοκρατική Ευρώπη δεν φοβάται όλους αυτούς που υπηρετούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βόζεμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στόχος εγκληματιών που εκτός των άλλων δρούν μέσω του διαδικτύου, δεδομένου ότι είναι στη χρήση τους το ανώνυμο διαδίκτυο, το διαδίκτυο στο οποίο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η ιδιότητα των ιδιοκτητών. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε πλημελήματα του κοινού ποινικού δικαίου όπως η απειλή ή η εξύβριση, αναφέρομαι στο οργανωμένο έγκλημα στο οποίο εντάσσονται κακουργήματα του τύπου εμπόριο ανθρώπων, οργάνων, όπλων, η παιδοφιλία, σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Τίθεται, όπω γνωρίζετε, σε κίνδυνο η ζωή και οι ελευθερίε των θυμάτων, αλλά και η κοινωνική ασφάλεια, η οικονομία και η καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Η αντιμετώπιση, κύριε Επίτροπε, είναι άνηση και τούτο γιατί οι συγκεκριμένοι εγκληματίες διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία που στην πλειονότητά τους οι διοκτικέ αρχές υστερούν πιστεύετε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η νομοθεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που διασυνοριακά τελείται μέσω του διαδικτύου καθώς επίσης και οι τρόποι δράσης και συνεργασίας των αστυνομικών αρχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι διασυνοριακό μόνο το πρόβλημα. Έτσι όπως εξελίχθηκε έχει πάρει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις. Εμάς η βασική μας στόχευση είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ασφαλούς ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι μια μεγάλη κατάκτηση μέσω της τεχνολογίας, της γνώσης και της ενημέρωσης και της καλύτερης επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Βέβαια, έχει γίνει abusement. Έχει γίνει κατάχρηση αυτής της ε, δυνατότητας που θέτει όλους μας πρώτης ευθύνης να προστατεύσουμε κυρίως τα θύματα. Και θύματα είναι πολλά. Θύματα είναι τα παιδιά, θύματα ε, ναι, είναι ε, όλοι αυτοί που την χάνουν εκμετάλλευση, είναι ο διασυρμός, είναι η αποκάλυψη προσωπικών ε, δεδομένων, είναι η πρόθεση μέσα από εκεί της ε, διαφθοράς. Είναι έγκλημα και όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί, ότι είναι και εσείς είστε διακεκριμένοι ποινικολόγος και το ξέρετε έγκλημα offline είναι και έγκλημα online. Υπάρχει όμως πολιτική. Υπάρχει η Budapest Convention on Cybercrime. Το κυβερνοέγκλημα έχει αρχίσει να μας απασχολεί πάρα πολύ και μόνο εμάς. Όλο τον κόσμο. Τον απλό πολίτη στην καθημερινότητά του. Εγώ πιστεύω ότι μιας και είναι ένα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιο ε, που εφόσον και συγκρίνεται μου ανατεθεί θα είναι υψηλή προτεραιότητα. Και αυτό θα γίνει στη συνεργασία μαζί σα και πάντοτε υπό την βασική αυτή προπόθεση που θέτω και το επαναλαμβάνω κουραστικά, χωρί να φύγετε σε τίποτα το πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων και τη αρχή αναλογικότητα. Και αυτή την την προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί πολλέ φορέ λειτουργούμε ασύμετρα. Δηλαδή περισσότερα μέτρα με λιγότερε επιπτώσει και συνέπειε ή και το ανάποδο. Σα ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ κυρία Τάνια Φαϊόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο κύριε Προτινόμενα Επίτροπε. Μιλήσατε ήδη για τα έξυπνα τα ευφύη σύνορα, smart borders. Ερωτώ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξέφρασαν κάποια προσδοκία ώστε στα μέσα 2016 να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πακέτο αυτό. Και εσείς ως Επίτροπος θα προτείνετε αλλαγές στο προτινόμενο πακέτο. Γιατί είχαμε πολύ σοβαρούς δισταγμούς και επιφυλάξεις στο Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά, της διατήρησης των δεδομένων, της αναλογικότητας, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και ως προς το ύψος των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για την ε, διεξαγωγή ελέγχων. Γιατί απαιτούνται πολύ περισσότερα κονδύλια για, ελέγχους αυτούς, για τους ελέγχους αυτούς. Ακούσαμε πρόσφατα ε, τις επικρίσεις για το υψηλό κόστος του δεύτερου συστήματος πληροφοριών Σέγγεν και στα τέλη του έτους ε, θα έχουμε κάποια ανάλυση για τα διαφορετικά, ε, διαφορετικές δυνατότητες του πλωτικού προγράμματος. Πώς αντιδράσετε. Ε, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι στις αρχές του 2015 θα, ναι, θα προχωρήσουμε σε ε, αναθεώρηση της, ε, της πρότασης. Υπάρχει και μία μελέτη που όπως ξέρετε είναι σε εξέλιξη και πιστεύω σύντομα να είναι στα χέρια της Επιτροπής. Ε, και ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου, ειδικότερα για το θέμα των smart borders. Και εύλογα το Κοινοβούλιο έχει προβάλει θέσει επιφυλάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αναφερικά με, με την αρχή τη αναλογικότητα και των ε, ε, fundamental και των ε, ε θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει όμω και κάτι άλλο. Το υπενηχθήκατε. Το κόστο. Είπα πριν και το επαναλαμβάνω και τώρα, η υπόθεση του SIS είναι ένα πολύ καλό μάθημα που πήραμε. Και γι' αυτό το λόγο η μελέτη που θα γίνει πρέπει να προβλέψει ώστε να μην οδηγηθούμε σε υπερβολικές δαπάνες που δεν θα αναλογούν στις πραγματικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, περίπου 500 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτονται την Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις λένε ότι μέχρι το 2020 θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για την σωστότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων ένα σύγχρονο σύστημα που θα στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες οι οποίες πάντοτε και το επαναλαμβάνω θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλίζουν τα ατομικά δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το privacy που είναι πολύ σημαντικό και βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Διότι όπως είπαμε, και καλά κάνατε και μου το θυμήσατε, η υπόθεση της Σέγγεν είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Thank you for that comprehensive... Ευχαριστώ για αυτή την ε, ε, συνολική απάντηση. Η κυρία Τερέζα Χιμένης Μπουσερίλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βραμόπουλε. Το πρόγραμμα της Σοχόλμης εγγυάται μια Ευρώπη ανοιχτή και ασφαλή, αλλά οι πολίτες μας αρχίζουν να αμφιβάλλουν ότι μπορούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους σε ό,τι αφορά μια τρομοκρατική επίθεση. Τι ε, σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μέτρα να λάβει για να αποτρέψει πιθανές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις από τους ξένους μαχητές στο Ιράκ και στη Συρία. Αυτοί οι μοναχικοί λύκοι όπως ονομάζονται που επιστρέφουν στην Ευρώπη και πώς θα αποτρέψετε τη στρατολόγηση των νέων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ε, πάνε στο τζιχάτ. Και σε σχέση με την τρομοκρατία θα ήθελα να γνωρίσω ποια είναι η πρόθεσή σας για τα θύματα της τρομοκρατίας. Ως Επίτροπος θα έχετε την απαραίτητη ευαισθησία προς τα θύματα της τρομοκρατίας, δίνοντα ιδιαίτερη προσοχή, υποστήριξη, προστασία και αναγνώριση, κοινωνική αναγνώριση που χρειάζονται για να εξομαλυνθεί η ζωή τους. Θα πάτε πιο πέρα από το πακέτο για τα θύματα με νομοθετική πρωτοβουλία ειδικό μέσο για τα θύματα ειδικά της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας, σας ευχαριστώ. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα και ξεκινώ ίσως από την πιο ευαίσθητη πτυχή του που είναι τα θύματα. Δεν θα πω κάτι κοινότυπο. Το ίδιο θα απαντούσε ο καθένας από εσά αν ήταν στη θέση μου. Αξίζουν και έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας. Γνωρίζετε ότι έχουμε ε, θεσπίσει και η μέρα θυμάτων ε, τρομοκρατίας ε, στην Ευρώπη. Αλλά, αν να πω, οι αρχές αυτές να μην είναι σλόγγαν πρέπει να είναι πολιτικές. Γι' αυτό απαντώ και στο άλλο σκέλος της παρατήρησής σας για το αν χρειάζεται μια νέα νομοθεσία. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Διότι θα πρέπει να το δούμε και αυτό ολιστικά. Οι foreign fighters είναι μια νέα πραγματικότητα, μιλήσαμε γι' αυτό πρωτήτερα. Και βέβαια πρέπει να προωθούν το συντομότερο ειδών συνεργασίε ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη με συντονιστικέ και υποστηρικτικέ υπηρεσίε από εμά για να μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Υπάρχει ανάγκη να δίνουμε έμφαση στην ε, ανταλλαγή ε, πληροφοριών και βέβαια να μην ξεχνάμε και την άλλη υποχρέωσή μας που πρέπει να αποτελέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που σε κάποια στιγμή πρέπει εμείς να εικονίσουμε και νομίζω θα αποτελέσει ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσουν για το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί και να χτυπηθεί ο φονταμενταλισμός και ο ριζοσπαστισμός στην πηγή, στη βάση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και όπως πολύ σωστά περιγράψετε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί μια ασύμετρη απειλή μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες μας. Και όσο και αν καμιά φορά αυτά τα δύο θέματα που αφορούν τους πυλώνες του χαρτοφυλακίου μπορεί να βρίσκονται και σε αντίφαση μεταξύ τους, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τον παράγοντα ασφάλεια. Θέλουμε μια ασφαλή Ευρώπη υπό την έννοια ότι οι πολίτες αυτής της νέας μεγάλης μας χώρας να αισθάνονται ασφαλείς στο έδαφό τους για να μπορούν να προωθήσουν τα όνειρά τους και τις επιδιώξεις τους μέσα σε περιβάλλον δημοκρατίας και ελευθερίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ηλιάνα Ιώτοβα, που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ, κύριε Κλοντ. Κύριε Αβραμόπουλε, έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πώς ε, θα μεριμνήσετε ώστε να γίνει σεβαστός ο κώδικας Σέγγεν μετά την πρόσφατη πρόταση για την επανεισαγωγή των ε, ελέγχων στα σύνορα. Δεύτερη ερώτηση. Θα ασκήσετε επίσης το Συμβούλιο ώστε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν. Γνωρίζετε το θέμα αυτό. Ε, και είναι ένα θέμα που απασχολεί και τα κρατη και το Συμβούλιο εδώ και μια τετραετία. Πρέπει να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί. Δεν αποδέχομαι προτάσεις που αποβλέπουν στον περιορισμό της ζώνης Σέγγεν. Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα από τι γράφεται και ακούγεται, Σέγγεν είναι μία από τις, το είπαμε και πρωτήτερα, μεγαλύτερες κατακτήσεις. Πρέπει πάση θυσία να το διαφυλάξουμε αυτό που είναι κοινή μας κατάκτηση και να το προστατεύσουμε. Σέγγεν με το πλέγμα αρχών που συνοδεύουν αυτήν την τόσο σημαντική απόφαση διασφαλίζει το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη μετακίνηση. Συνεπώς δεν τίθεται τέτοιο θέμα και επιτρέψτε να πω και όσοι το επαναφέρουν καμιά φορά να ξέρουν ότι δεν συμβάλλουν σε αυτό για το οποίο όλοι βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή, δηλαδή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ξέρετε, στην ευρωπαϊκή διαδικασία δύσκολα οδηγούμεθα σε κατακτήσεις. Πρέπει να φέρουμε κοντά αντίθετες απόψεις, συγκρουόμενα συμφέροντα, εθνικές απόψεις. Το ότι καταφέραμε να κάνουμε κάτι και το προστατεύουμε, αυτό λυπάμαι πρέπει να είναι έξω από κάθε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δική μου θέση εάν και εφόσον αναλάβω αυτά τα καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλο τη ερώτησή εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο για τη Βουλγαρία η τη Ρουμανία, δύο χώρε που γνωρίζω επίση πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό ξεφεύγει από τη δική μου άποψη, γιατί είναι γειτονικέ χώρε, την χώρα που με ξέρει και την ξέρω καλύτερα, αλλά πλήρουν πλήρω τι προποθέσει. Ναι, δεσμεύομαι ότι συντομότατα και οι δύο αυτέ χώρε θα αποτελούν μέρο τη οικογένεια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, εγώ θα αναφερθώ στη μελλοντική πολιτική θεωρήσεων διαβατηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα ε, είχε μια φιλελεύθερη ε, πολιτική και κάθε απελευθέρωση θεώρησης έρχεται πάντα σε σύγκρουση, σε ένταση με τις αυξαμένες απαιτήσει για την εσωτερική ασφάλεια. Ας πούμε, οι περισσότεροι παρανόμως διαβιώνται στην Ένωση έρχονται νόμιμα, αλλά παραμένουν ε, περισσότερο από όσο τους επιτρέπει η βίζα που έχουν. Ερωτώ λοιπόν, πώς ως αρμόδιος επίτροπος για την μετανάστευση αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών θα εξασφαλίσετε η εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιβαρυνθεί από μια πολύ πιο χαλαρή πολιτική για την θεώρηση διαβατηρίων και να μην καταργηθεί τελικά. Θα έχετε μια πιο ανοιχτή, πιο περιοριστική πολιτική. Και πώς βλέπετε το διάλογο που γίνεται με την Τουρκία για την απελευθέρωση θεώρησης και την πίεση ε, για τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Αφού σας ευχαριστήσω θα ήθελα να πω ότι ε, αυτό που λέμε case by case examination ε, ασφάλεια είναι μία από τις προϋποθέσεις, δηλαδή από τα ε, preconditions που υπάρχουν. Είναι αλήθεια επίσης και το υπενηχθήκατε με την ερώτησή ότι κάποιες χώρες δεν μπορούν ακόμα να, ε, να τους δώσουμε visa liberalization. Υπάρχουν κάποιες όροι, και κάποιες ε, προϋποθέσεις. Αλλά η visa policy έχει σε σκοπό να διευκολύνει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων από όλο τον κόσμο να μπορούν να επισκέπτονται την Ευρώπη. Μιλάμε για φοιτητέ. Φαντάζομαι και εσεί και εγώ περίπου τη ίδια ηλικία είμαστε. Κάποτε ταξιδεύαμε από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη και αυτό ήταν δύσκολο την εποχή εκείνη. Πρέπει να διευκολύνουμε του νέου ανθρώπου να γνωρίζουν καλύτερα του άλλου ε, λαού. Εκεί δεν είναι θέμα διευκόλυνση, είναι θέμα βέβαια κάποιων όρων και κάποιων προϋποθέσεων. Η ερώτηση, η ερώτησή σας αν θα είναι πιο σφιχτή η πιο ανοιχτή πολιτική με οδηγεί στο να σας πω ότι θα πρέπει να είναι εκεί που πρέπει πιο ελαστική και εκεί που πρέπει βεβαίως πιο αυστηρή και ξέρουμε που πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Αλλά το να αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο σε ανθρώπους της δημιουργίας, της τέχνης, των γραμμάτων, των τεχνών και όλους αυτούς που συμβάλλουν στο πέρασμα του χρόνου στο να γίνεται πιο συνεκτική η Ευρώπη και ο κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Και το λέω γιατί είναι ίσω περιπτώ για την κουβέντα, αλλά όταν έκανα το πρώτο μου ταξίδι 19 χρόνων φοιτητή στην Ευρώπη, αναγκάστηκα να αλλάξω διαβατήριο στο Λονδίνο, γιατί είχε γεμίσει από τι φραγίδες το πρώτο που είχα πάρει μαζί μου και έπρεπε να το ανανεώσω πριν ακόμα λήξει. Αυτά είναι κατακτήσει τη γενιά μα που δούλεψε και δουλεύει για μια Ευρώπη ανοιχτή. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, Τουρκία. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει επικυρωθεί το, συγνώμη, Admission Agreement. Ο διάλογος για το Visa Liberalization ε, θα συνεχιστεί. Έχει αρχίσει. Και προτίθεμαι, ναι, να τον συνεχίσω όταν όμως αυτός γίνει ε, confirmed. Κυρία Καταρίνα Κινίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προτινόμενα Επίτροπε, μιλήσαμε για τις δεσμεύσεις που αναλάβατε σήμερα. Δέσμευση για να έχουμε πιο αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των λαθρέων διακινητών ή των εμπόρων ανθρώπων. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν αυτές τις μορφές εγκληματικότητας, τι συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβετε και σε νομοθετικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πώς θα προστατεύσουμε τους πολυάριθμους επίσης ασυνόδευτους ε, ανηλίκους. Γιατί αυτοί οι ανήλικοι είναι οι πιο ευάλωτοι και χρήζουν περισσότερης προστασίας από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες και αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Και αυτοί οι ανήλικοι στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τις εγκληματικές οργανώσεις για πορνή ανηλίκων ή για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ευχαριστώ. Ε, Τσινίτσι. Η ερώτησή σας είναι υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και θα σας απαντήσω ευθέως. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε να πω στα αγγλικά είναι τα τρία eyes στα αγγλικά, δηλαδή έρευνα, πληροφορίες, συγκέντρωση πληροφοριών και διεθνή συνεργασία. Υγείας κατευθύνσεις εν ώψη του 2015 που θα παρουσιάσω σε εσά, βεβαίω εάν είμαι εδώ σε αυτή τη θέση, ε, τη σχετική στρατηγική. Δεν θα μιλήσω για το τράφικινγκ, Ακούστηκαν τόσα πολλά σε αυτή την αίθουσα και νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα, ούτε μία από του συναδέλφου σα που δεν συμφωνεί με την άποψη. Απεινή πόλεμο και καταπολέμηση και των σμάγκλερ και των τράφικερ. Για τα παιδιά μα. Το πιο ευαίσθητο κομμάτι τη κοινωνία. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα ε, action plan το οποίο όμω τελειώνει αν δεν κάνω λάθο, τον επόμενο χρόνο. Εμεί εδώ, σε συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι θα είστε από τους πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοβουλίας, θα εκπονήσουμε ένα νέο σχέδιο δράσης. Με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το προηγούμενο, καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν και γενόμενοι στην πράξη πολύ πιο αυστηροί, πολύ πιο αποτελεσματικοί και βεβαίως παραμένοντας το ίδιο ευαίσθητοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Φρανκ Έγγελ, παρακαλώ. Κύριε Προτινόμενη Επίτροπε, στην εισαγωγή σας μιλήσατε για την ανάγκη να αποτρέψουμε να γίνει Ευρώπη φρούριο. Και συμφωνώ και με τα όσα είπατε για το Σέγγεν. Και σημειώνω ότι Πραγματικά εσείς ε, θα υπερασπιστείτε την ελεύθερη κυκλοφορία ε, στο χώρο Σέγγεν που είναι από τα μείζωνα επιτεύγματα και τις κατακτήσεις είπατε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα προσωπικά θα αγωνιστείτε γι' αυτό. Αλλά αν θέλουμε ε, και ο κόσμος και οι πολίτες που κατοικούν σε αυτή τη τεράστια έκθεση έχουν την αίσθηση ότι αποδίδει αυτό και έχει αποτελέσματα, δεν θα πρέπει από κοινού να φροντίσουμε τα εξωτερικά σύνορα να γίνουν τα ουσιαστικά κοινά ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Δηλαδή τελικά να καταφέρουμε να τα δεχειριστούμε με τρόπο τολμώ να πω ομοσπονδιακό, εν πάση περιπτώσει κοινοτικό, έτσι ώστε συνειδητά τα ελληνικά σύνορα να θεωρούν οι Λουξεμβούργοι συμπατριώτες μου ότι είναι και αυτά τα σύνορα του Σέγγεν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Έγγελ. Τώρα με στο να μιλήσω και λίγο πιο προσωπικά. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια ήμουνα ε, μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κινήματος και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Υπό την έννοια ότι πάντα πίστευα σε μια ενωμένη, ενιαία Ευρώπη, πολύ κοντά στο όραμα εκείνο που το δημιούργησα. Αλλά αυτό έχει σχετική αξία, ίσως περισσότερο για την καλύτερη γνωριμία μεταξύ μας. Αλλά ναι, συμφωνώ μαζί σας, ότι ο στόχος πρέπει να είναι μια μέρα να φτάσουμε σε αυτό που ήταν και το όραμα εκείνο. Τα ξεκινά εξωτερικά σύνορα, με κοινού κανόνε και χωρί ιδιαιτερότητε που να έχουν να κάνουν με εθνικέ ευαισθησίε. Ο δρόμος όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι μακρύ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ηλικία, αλλά θα το ζήσει η δική μα γενιά που το οραματίστηκε. Όταν έχουμε ασφαλή σύνορα, έχουμε εκ των πραγμάτων και μια ασφαλή ζώνη Σέγγεν. Δεν θα επανέλθω σε αυτό που πρωτήτερα, μου το θυμίσατε κι εσείς. Είναι η μεγαλύτερη για μένα κατάκτηση και η πιο χειροπιαστή στην πράξη. Ας την προστατεύσουμε, ας την ενισχύσουμε και μέσα από εκεί ας καλλιεργήσουμε περισσότερο την κοινή ευρωπαϊκή μας συνείδηση, πάντοτε στεκόμαστε με υπερηφάνεια στην καταγωγή μας, στην ιστορία των λαών μας και στις πατρίδες μας. Αλλά το μέλλον είναι η ενιαία Ευρώπη μέσα από κοινά σύνορα που όμως θα, έχει, θα συμπεριλαμβάνει και μια σειρά από κοινέ πολιτικές ευρωπαϊκής ενόρασης. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η Άννα Κύριε Αβραμόπουλα δεδομένη τη πρώτη έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Διαφθορά που δημοσιεύθηκε σε αρχέ του έτου και των νέων κανόνων για την πάταξη τη νομοποίηση όδων από παράνομε δραστηριότητε που θα περάσουν σε διαδικασία συνδιαλλαγή. Θα προτείνετε και άλλα μέτρα για να αντιμετωπίσετε τα συναφή προβλήματα τη διαφθορά, τη εισαφοροδιαφυγής και τη ε, νομοποίηση όδων από παράνομε δραστηριότητε. Επίσης θέλετε, θα, μπορούμε να έχουμε ένα δημόσιο προσιτό μητρό όλων των και των τραστ και άλλων ενδιαφερομένων σε στις, στις, στους τριμερείς διαλόγους και προτείνε, θα προτείνετε μια στρατηγική για να πατάξετε την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη αλλά και στη σχέση της με τρίτες χώρες και φορολογικούς παραδείσους. Σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό θα ήταν ένα τέτοιο publicly accessible register. Αυτό εννοούσατε φαντάζομαι με την, με την ερώτησή σας. Μην βιαστούμε. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Σίγουρα το ξέπλυμα, thank you Σίγουρα το ξέπλυμα του χρήματος, η κυκλοφορία μαύρου χρήματος, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά είναι υπαρκτά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με, με αποτελεσματικότητα. Κοινό στόχο μα είναι να βρούμε μεθόδου και τρόπου. Και ένα από αυτού ενδεχομένω να είναι αυτό που προτείνεται και το οποίο συγκράτησε. Η διαφάνεια είναι μια βασική αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά, γιατί όλοι διαβάζουμε εφημερίδε, παρακολουθούμε τι γίνεται στον κόσμο, η διαφθορά δεν έχει σύνορα. Συνηθίζω να λέω ότι δεν είναι η εξουσία που είναι διεφθαρμένη, αλλά η άνθρωποι που διαφθείρουν την εξουσία και τους μηχανισμούς. Επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής, σε κάθε τι που μπορεί να τον οδηγήσει σε τον δρόμο θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε συνολικά την κοινωνία, το σύστημα, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία. Ζητάμε επενδύσεις στην Ευρώπη. Και πολλές φορές οι επενδυτές βρίσκονται μπροστά σε ένα τείχος γραφειοκρατίας η οποία εκολάπτει και την αδιαφάνεια μέσα στις διοικήσεις. Βέβαια, για να μην ξεφύγω από το σκοπό αυτής της συνάντησης και από τα πλαίσια των δικών μου αρμοδιοτήτων εφόσον θεωρηθεί εκλεγώ ή γίνω, ε, εγκριθώ να είμαι ε, commissioner του χώρου, δεν είναι αποκλειστικά δική μου αρμοδιότητας. Προτίθεμαι όμως να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους μου κομισάριους, έτσι ώστε η μάχη κατά της διαφθοράς να αποδώσει και να είναι μία από τις υπερηφάνειες και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για την πενταετία που έρχεται. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί και τη θέληση έχουμε και τις ιδέες και τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Κυρία Χολμάγερ, ακούσαμε και συζητήσαμε πολλά θέματα για το θέμα των προσφύγων. Η κοινή γνώμη έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα για τους αριθμούς. Οι χώρες ε, όπως το Βέλγιο, η Μάλτα, η ε, Σουηδία και η Γερμανία είναι αυτές που δέχονται τους περισσότερους. Ε, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έρχονται να προσθεθούν, αλλά στην κοινή γνώμη υπάρχει στρεβλή εικόνα για το ποιος υποδέχεται και ποιους. τώρα, σε σχέση με τη σημερινή κρίση, στο νέο κανονισμό Δουβλίνου ε, ε, υπάρχει ένας μηχανισμός για την ε, έγκαιρη προειδοποίηση, για την αντιμετώπιση και αποφυγή των κρίσεων. Θα φροντίσετε επιτέλους να υπάρξει ένας συντονισμός, μια συνεργασία με το των μελών, για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και με το ΕΑΣΟ και όλα τα άλλα που υπάρχουν ως δυνατότητες, περισσότερο από ό,τι γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χολμάγερ. ναι, το άρθρο 33 στο Δουβλίνο είναι σαφές. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις για να πετύχει. Αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη. Αυτό δοκιμάζεται καθημερινά ε, στην πράξη. Και προς αυτή την κατεύθυνση, κατά την γνώμη μου, πρέπει να κινηθούμε. Συμμερίζομαι και την παρατήρηση που κάνατε για την ανησυχία των πολιτών. Διότι αυτή είναι οι αποδέκτες της δικής μας πολιτικής. Καμιά φορά, ξέρετε, σε αυτούς τους χώρους ακούγονται πολύ ωραία συνθήματα. Εγώ θα τελειώσω, θα κλείσω μάλλον την απάντησή μου με μια πολύ απλή επισήμαση όπως ακριβώς μου έρχεται. Η solidarity να πάψει να είναι σλόγγαν και να γίνει πολιτική στην πράξη και συνείδηση όλων των κρατών μελών. Και τότε οι πολίτε που σα επεσήμαναν αυτά τα πράγματα θα έρθουν και θα σα πούν ότι επιτέλου ζούμε σε μια αλληλέγγυα Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πίτερ Νίντε Μίλλερ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Οριστέντα, Επίτροπε, η στρατηγική εδώ είμαι, για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης ε, μπαίνει σε μια νέα περίοδο, μια νέα πενταετία και χρειάζεται συντονισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης σε συνεργασία με τρίτες χώρες σε θέματα καλύτερης ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί και νέες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας. Οι δικές σας προτεραιότητες ποιες είναι για το επόμενο διάστημα, για την εσωτερική ασφάλεια και τη στρατηγική αυτή και θα δεσμευτείτε ότι θα αξιοποιήσετε πλήρως και θα εξαντλήσετε τα υφιστάμενα μέσα στην Ένωση για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και σοβαρού εγκλήματος και τις συμφωνίες αμοιβαία νομικής συνδρομής για αστυνομική και δικαστική συνεργασία πριν έρχεται τώρα να δημιουργείτε καινούρια μέσα. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δημιουργήσουμε καινούργια μέσα. Έχουμε τα μέσα, έχουμε τις δυνατότητες, πάνω απ' όλα έχουμε την πολιτική ε, βούληση. Απαντώ ευθέω στο ερώτημά σα. Δεν χρειάζονται καινούργιοι θεσμοί, χρειάζεται όμω μια καινούργια security policy. Ε, μια καινούργια security strategy, θα έλεγα. Πάνω στι αρχέ βέβαια που επανειλημμένα ε, θίξαμε και αναφέραμε κατά τη διάρκεια τη σημερινή συνάντηση, δηλαδή σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της παρατομικών ε, ελευθεριών και τη αρχή αναλογία. Ε, μου επιτρέψετε πάλι να πω κάτι όπως αυτές τις, το τον καιρό, μελετώντας ε, τα θέματα αυτά, για παντός στο ερώτημά σα, διότι τι προτίθεται να κάνουμε. Είναι ένα P και τρία I's, όπω λέει. Το P είναι protection. Τα I's είναι information, innovation και πάλι international cooperation. Διότι όλα αυτά που λέμε, αν υπάρχει διεθνή συνεργασία, δεν θα αποδώσουν και θα είναι απρόσφορες και αναποτελεσματικές οι πολιτικές. Νέα όργανα δεν θα διαφωνήσω μαζί σα. Ίσως να μην χρειάζονται. Νέες μέθοδοι όμως χρειάζονται. Νέα συστήματα υποστηρικτικά και από τις νέες τεχνολογίες και κυρίως από αυτό που σας είπα πρωτήτερα από μια στενή αλληλέγγυα συνεργασία. Είναι μια, αν θέλετε, άποψη επί της αρχής, αλλά που νομίζω είναι πολύ κοντά και στο πνεύμα της ερώτησής σας, αν καλώς το ερμήνευσα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση, παριθμό 45 από τον κύριο Εμίλ Ράντεφ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε προτινόμενε επίτροπε. Το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και η διαφθορά είναι παγκόσμια φαινόμενα και απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις. Άρα χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα ε, βάσει προοδευτικών νόμων. Ε, την περασμένη θητεία συστήθηκε μια επιτροπή που εκπώνησε κάποιες συστάσεις ε, σχετικά. Για παράδειγμα, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων η διαφθορά, ας πούμε, θα πρέπει να είναι υψηλά στις προτεραιότητες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που δημεύονται και κατάσχονται για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος. Ε, τι προτίθεστε λοιπόν να κάνετε εσείς, ε, κινώντας από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λάβετε κάποια μέτρα. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη συνέχεια. Για την αστυνομική συνεργασία χρειάζεται και προβλέπεται περαιτέρω οικονομική ε, ενίσχυση. Έχει αποδώσει καπούς. Ξεκινώ από το τελευταίο, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που διατίθεται ε, εάν το ξοδέψουμε ορθολογικά θα αποδώσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ΚΡΙΜ. Έχει κάνει καλή δουλειά η ΚΡΙΜ. Η δε έκθεσή της, ε, πρέπει να σας πω ρίχνοντας μια ματιά, είναι εντυπωσιακή ως προς το περιεχόμενό της. Ο σκοπός ποιος είναι. Ο σκοπός είναι η πλήρης διάλυση, the dismantlement όλων, των οργανωμένων δικτύων καταπολέμησης. Και είναι ένας από τους σκοπούς που καλείται να υπηρετήσει η, Επιτροπή. Αλλά και αυτό πάντα σε συνεργασία μαζί σας. Ανάλογα λοιπόν με το assessment που γίνεται αυτή τη στιγμή, θα δω και τι πρωτοβουλίες θα αναλάβω. Θα ήταν πολύ πρόχειρο από μένα να κάνω ανακοινώσεις μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τα hints που κάνατε μέσα από την ερώτησή σας με οδηγούν σε ένα βαθύτερο προβληματισμό και θέλω να πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε μαζί την πρότασή μας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με όλες τις, αυτές τις παραμέτρους, τότε πραγματικά θα έχουμε κάνει σημαντικά ένα βήμα μπροστά. Πάντως, ένα πράγμα μας ενώνει, η απόφασή μας να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Και βεβαίως η ΚΡΙΜ, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ακούγεται πάρα πολύ η, η δουλειά που κάνει, έχει κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά την οποία οφείλουμε και να τις αναγνωρίσουμε. Κύριε Προτινόμενο Επίτροπε, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ε, για αυτή τη μαραθώνια συνεδρίαση. Φυσικά ήταν πολύ έμπειρα με εξοικειωμένα με το θέμα και θα συμφωνείτε ε, κύριε Επιτροπέ ότι αυτή είναι μία από τις πέντε ακροάσεις που συμμετέχουμε αλλά πραγματικά βρίσκεται στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων μας το θέμα της μετανάστευσης του ασύλου, της ε, παράτυπης μετανάστευσης είναι από τα πιο σημαντικά θέματα για μας και γι' αυτό οι συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι και ενέκυψα ε, στις λεπτομέρειες του θέματος. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ και τον προτινόμενο Επίτροπο για την προετοιμασία του για την ακρόαση αυτή. Δεν θα προδικάσω, θα, θα προεξοφλήσω τις περαιτέρω δράσεις, γιατί εναπόκειται στα μέλη της Επιτροπής μέσω των συντονιστών να κρίνουν αυτά που είπατε σήμερα. Και μάλιστα η συνεδρία θα γίνει στις 5 η συνεδρία των συντονιστών για την αξιολόγησή σα. Θα ήθελα εγκατακλείδη να σταθώ σε μερικά πράγματα που είπατε. Αναλάβατε τη δέσμευση να αναθεωρήσετε του μηχανισμού για την λαθρομετανάστευση και τον το σχέδιο της οριζόντιας νομοθεσίας, καθώς θα κάνετε μία ανάλυση της οδηγίας για την κράτηση δεδομένων μετά την πρόσφατη νομολόγια του ΔΕΚ. Επίσης, μιλήσετε για μία ενημερωμένη πρόταση για τους φαγγέλους επιβατών, ώστε να ε, γίνονται σεβαστές ε, οι αρχές προστασίας δεδομένων. Επίσης, μιλήσετε για τις πρωτοβουλίες της Frontex. Πιστεύω ότι απαντήσατε σήμερα σε σημαντικές προτάσεις και των μελών της Επιτροπής μας, αλλά φυσικά εμείς ε, θα αξιολογήσουμε τη σημερινή ακρόαση με βάση τις ικανότητές σας και με βάση αυτά που μας είπατε σήμερα. Επαναλαμβάνω, η συνεδρία αξιολόγηση θα ξεκινήσει στις 5. Μπορεί να έμειναν κάποιες ε, ερωτήσεις αναπάντητες. Ε, θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον προτινόμενο επίτροπο για τελικά σχόλια. Τρία λεπτά. Αν επεκταθεί στα πέντε λεπτά θα χάσει όλη την υποστήριξη που κέρδισε νωρίτερα στο κρατήριο. Αν κάνετε κατάχρηση του χρόνου σας θα αποφασίσετε, αλλά ελπίζω να, λάβατε το, να καταλάβατε το υπονοούμενο. Τρία λεπτά είναι αρκετά γιατί είμαστε όλοι εξουθενωμένοι. Τρία λεπτά παρακαλώ για να ολοκληρώσετε και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Προτινόμενο Επίτροπε, σας ακούμε για τα τελικά σχόλια και σας ευχαριστώ και πάλι. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πραγματικά με διαφωτίσατε σε πολλά θέματα για τα πολύ ευαίσθητα αυτά ζητήματα φεύγω από την αίθουσα πιο εμπνευσμένο, πιο ενθαρρυμένο για τα νέα μου καθήκοντα, εφόσον φυσικά ε, επιβεβαιώσετε ως Επίτροπο και αν τελικά επιβεβαιωθεί η υποψηφιότητά μου θα είμαι ο πρώτος Επίτροπος ε, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τέτοιο θα επικεντρώσω την πολιτική μου πείρα σε τρεις άξονες δράσης. Καταρχήν θα προσπαθήσω να διασφαλίσω, όπως προτείνατε κι εσείς, ε, να εγκρίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ολιστική, σφαιρική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική που θα στηρίζεται στις αρχές της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης, αλλά φυσικά και στην ευθύνη. Επίσης θα αντιμετωπίσω κάποιες σημαντικές προκλήσεις στην ασφάλεια εν των νέων απειλών και των νέων προκλήσεων με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και έχοντα επίγνωση τη ευθύνη ε, τη εξασφάλιση ε, ενό προστατευμένου και ασφαλού περιβάλλοντος για του πολίτες. Επίσης ε, θα συνεχίσω στην πολιτική εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευση σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να έχουμε έναν διαφανή, ειλικρινή και συνεχή διάλογο μεταξύ μας. Θα συνεργαστώ μαζί σας με βάση τη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Thank you. Thank you. Εμείς σας ευχαριστούμε. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστούμε κύριε Προτινόμενη Επίτροπε. Ακολουθήσατε τη συμβουλή μου. Λήξη στις ακροάσεις.